Αγαπητοί συνάδελφοι, ας βρει καθένα στη θέση του όπως νομίζει σε αυτήν την πρωτότυπη αίθουσα. Αυτή είναι και η γοητεία των κτηρίων στις Βρυξέλλες, χωρίς άλλα σχόλια. Και επειδή οι πρώτοι μας ομιλητές είναι εδώ, μπορούμε να αρχίσουμε. Στο σημείο 1, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, προτείνω να αλλάξουμε τα σημεία 3 με, το σημείο 3 με το σημείο 6. Αν δεν έχετε αντίρρηση, πάμε στις ανακοινώσεις, έχω να κάνω τρεις. Πρώτη, για την έκθεση Θέρκας σχετικά με τις αναδιαρθώσεις θέλετε να έχουμε, στην... θα το συζητήσουμε στους συντονιστές, αλλά θέλετε να συζητήσουμε και στην Ολομέλεια της Επιτροπής ε, τις ε, μελέτες της ομάδας των εμπειρογνωμόνων για την προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό θα μπορούσε να γίνει στις 9 Οκτωβρίου. Αυτό θα μας οδηγούσε βέβαια στην αναβολή της ψηφοφορίας της έκθεσης Θέρκα σε μια έκτακτη συνεδρίαση τον Νοέμβριο. Σημείο Β. Αναμεταδίδεται η συνεδρίαση μέσω του διαδικτύου. Τρίτον, και έπρεπε να είχα ξεκινήσει από αυτό γιατί είναι το πιο ευχάριστο, αύριο προτείνω να αποχαιρετήσουμε την ε, υπάλληλου της Επιτροπής, την κυρία Μποζίτσα, η οποία μας εγκαταλείπει για μια άλλη Επιτροπή. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι έχετε κέφι. Κοιτάστε, είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο να μιλάτε πίσω από την πλάτη μου, λοιπόν, με ενοχλείτε. Πάμε στο σημείο 6 και δίνω το λόγο στον Τόμας Μαν για να μας παρουσιάσει για να μας παρουσιάσει την έκθεση που σας μοιράστηκε. Τις συμβαστικές τροπολογίες είναι υπηρεσίες εδάφους στα αεροδρόμια της Ένωσης. Πρόκειται για ένα κείμενο για το οποίο πρέπει να ψηφίσουμε αύριο. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβουργό είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις. Ε, μερικές εξ αυτών ήταν διμερείς και είχαμε και μια κοινή συνάντηση. Προέκυψε λοιπόν από τις συναντήσεις αυτές ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στο ανώτατο όριο, ε, δηλαδή ε, τέτοιο το θέμα κατά πόσο μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα που να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και συμβιβαστική πρόταση. Όσον αφορά λοιπόν στις συμβαστικές προτάσεις, Πράγματι, κατορθώσαμε κάπου να καταλήξουμε. Βέβαια, κατά πόσον θα παραμείνει, θα εξακολουθεί να ισχύει ο συμβασμός. Ε, αυτό θα κριθεί και από τις συνεδριάσεις των παράλληλων ε, συνεδριάσεων ε, που λαμβάνουν χώρα. Πολιτικές ομάδες δεν συμμετείχαν. Οι πράσινοι είπαν ότι όσον αφορά στην πρόταση επιθυμούν να απορρίψουν ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σύνολο της πρότασης. Ε, βεβαίως ε, δεν ξέρω τι επιθυμούν οι πράσινοι αγνώντας αυτήν την ε, συμβαστική πρόταση που πετύχαμε με μεγάλη προσπάθεια. Και αν δεν καταλήξουμε τότε το αποτέλεσμα θα είναι ότι η Επιτροπή Μεταφορών θα είναι η μόνη υπεύθυνη και όλα αυτά που έχουμε επεξεργαστεί, δηλαδή δικαιώματα για τους εργαζομένους, η ε, μεταβίβαση διαφόρων επιχειρήσεων και τρίτο θέμα την εκπαίδευση. Όλα αυτά δεν θα μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε σε νέα έκθεση, διότι θα έχουμε αποσύρει την παράγραφο 50 που αφορά τις ε, ίδιες αρμοδιότητες Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει dumping μισθών, να μην χαθούν θέσεις εργασίας και νομίζω ότι βεβαίως θα ήταν καλύτερα να έχουμε προσφέροντες που να γνωρίζουμε ε, το τι μπορούν να μας εγγυηθούν. Και κάτι άλλο να πω. Υπάρχει στα αεροδρόμια υπάρχουν διάφορες συνθήκες. Δηλαδή δεν μπορεί να βρεθεί λύση για όλα δεν μπορούμε ε, να κάνουμε τίποτα. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι επιθυμούμε την προστασία των εργαζομένων. Τα θέματα που αντιμετωπίζουμε διαφορετικά είναι τα εξή. Για ποιου τομεί θα ισχύουν όλα αυτά και εγώ τίνω να συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δηλαδή μπορούμε να επεξεργαζόμαστε μόνο θέματα ε, στα οποία είναι περιορισμένος ο ανταγωνισμός. Ε, βεβαίως ε, στη συμβαστική πρόταση λέμε ότι καλούμε τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν κατά πόσον πέρα από αυτούς τους ε, τέσσερις τομείς είναι δυνατόν να εξεταστούν και άλλοι. Με άλλα λόγια, το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των κρατών μελών. Τώρα, όσον αφορά την ε, διατήρηση θέση εργασίας ε, σε περίπτωση εξαγοράς της ε, εταιρεία, μέχρι τώρα υπήρχε η δυνατότητα απόλυση εργαζομένων. Εμείς, για καθαρά οργανωτικούς λόγους, καταλήξαμε σε μια πολύ καλή σημαστική πρόταση. Η Α είναι και ο πυρήνα των προσπαθειών μας. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν και ισχυρότερε εγγυήσεις, αυτό στο ΑΒ. Υπάρχουν και άλλε συμβαστικές προτάσεις που τι θεωρώ πολύ σημαντικέ, όπω παραδείγματο χάνει η ΣΥ όπου είναι απαραίτητο καταρχήν οι εργαζόμενοι να έχουν το δικαίωμα να ε, μπορούν να διαβάσουν την, ε, ε, τις προδιαγραφές που θα ισχύουν μετά την εξαγορά της επιχείρησης. Αυτό που επίσης βρίσκουμε σημαντικό είναι στο ΔΕΛΤΑ οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι προφανώς και να απασχολούνται, αλλά ο έλεγχος θα πρέπει να παραμένει στις αρμόδιες αρχές. Δηλαδή όχι μία αρχή, αλλά να μεριμνούμε έτσι, ακριβώς επειδή υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις στα κράτη-μέλη, να πούμε ότι οι προδιαγραφές για κάθε αερολιμένα θα πρέπει να την χάνει επεξεργασία από την αρμόδια αρχή σε συνεργασία με το φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου και με τους κοινωνικούς εταίρους. Όλα αυτά τα βρίσκω πολύ σημαντικά. Και κάτι άλλο, επειδή δεν μπορούμε να μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θέλω να επισημάνω ορισμένα θέματα. Τίθεται το ερώτημα, τι θα γίνει με τη διάρκεια εκπαίδευση. Υπάρχουν μερικοί που λένε η διάρκεια αυτή να είναι δύο ημέρες. Η Κομισιόν λέει αυτό αρκεί. αρκεί. Φτάνει και περισσεύει. Έχουμε όμως και ε, διαφορετικές, διαφορετική ποιότητα ε, παροχής πλαισιών. Όταν είναι πολύ καλή δεν αρκούν οι δύο ημέρες, γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε τουλάχιστον πέντε ημέρες εκπαίδευση. Και όσον αφορά στην ποιότητα, δηλαδή οι, τα, ε, δοκιμές, η εκπαίδευση, όλα αυτά θα πρέπει να εναρμονιστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο που ε, το κατά πόσον η εκπαίδευση είναι προσαρμοσμένη στην ποιότητα και η ερμηνεία του ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις και πώς ε, παραμένουν αξιοπρεπείς, αυτό ορίζεται από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να τα επανεξετάσουν όλα αυτά, γιατί εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει συνένεση για την κοινωνική Ευρώπη. Επ' αυτού εργαστήκαμε όλοι από κοινού. Ελπίζω λοιπόν οι συμβαστικές προτάσεις που κατατέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν και σήμερα και σε τελική ανάλυση να καταλήξουμε σε κάτι ε, το οποίο θα αποτελεί σαφές δείγμα για τους εργαζόμενους και όχι απλά έτσι μια πολύ φιλική ρήτρα ε, όπου να λέμε ότι εντάξει ας συμφωνήσουμε σε αυτό και μετά για yeah, του. το. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να διασφαλιστεί η κοινωνική Ευρώπη. Ευχαριστώ η Ιούτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινώ με το εξή. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένη με αυτά τα οποία επιτέχθηκαν στις ε, διαπραγματεύσεις. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξή ε, βλέποντας ε, και τις αντιδράσεις των πολιτικών ομάδων πριν από τη συνεδρίασή μας, αυτά τα οποία άκουσα πόρο απέχουν από αυτά που επιθυμούμε. Ο κύριος Μαν παρουσίασε μια κατάσταση την οποία αντιμετωπίζω και εγώ. Δηλαδή, αν καταψηφίσουμε την έκθεση, υπάρχει κίνδυνος οι εργαζόμενοι να απολαύουν μικρότερης ακόμα προστασίας από αυτήν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα των σοσιαλδημοκρατών προς όφελος των εργαζομένων θα αναγκαστεί να υπερψηφίσει. Ελπίζω βέβαια στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή σε μια μεταγενέστερη φάση να αποσυρθεί η πρόταση αυτή. Δεν είναι αλήθεια ότι εμείς ε, στην περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης μπορούμε να προστατεύσουμε μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν ισχύει αυτό. Και θέλω να πω ότι ε, όσον αφορά τους ε, συμβασμούς που επιτύχαμε, ξέρετε που θα καταλήξουμε, θα έχουμε εργαζομένους πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στις επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν μια ε, διατύπωση που τέλος πάντων ε, καλύτερα από το τίποτα, αλλά οι ε, περισσότεροι συμφωνούν ότι δυστυχώς δεν μπορούσε να εξευρεθεί άλλη λύση. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι να τηρούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Ήταν δύσκολο να το προσπαθήσω, να διατηρηθούν επίσης και οι ε, συνθήκες εργασίας στην περίπτωση υπεργολαβιών, ε, δύσκολη η συμβαστική πρόταση, καλύτερα βέβαια από αυτό που είχαμε παλαιότερα. Αυτό που χρειάζεται απαραίτητα είναι να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές για την περαιτέρω εκπαίδευση και την κατάρτιση. Και νομίζω ότι βεβαίως και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εθνικές ε, ιδιομορφίες που υπάρχουν σε κάποιους αερολιμένες. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η κοινωνική Ευρώπη Ευρώπη για τους εργαζόμενους. Μήπως είναι απλά κενά λόγια και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους από την πλήρη απελευθέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, για μας, ε, τους φιλελεύθερους, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι εμείς σαφώς και είμαστε υπέρ του μεγαλύτερου ανταγωνισμού και περισσότερης ε, απελευθέρωσης. Ε, Κατονούμε βέβαια το πρόβλημα. Εδώ πρόκειται για εργαζόμενους που βρίσκονται σε έναν τομέα με χαμηλούς μισθούς και οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πολλές από τις συμβαστικές προτάσεις τις απορρίπτουμε. Πολλές από αυτές ε, που κατέθεσε σήμερα ο συνάδελφος κύριος ε, Μαν. Ισχύει λοιπόν το εξής. Και να σας πω ε, το εξής, καθαρά στρατηγικά. Βεβαίως εδώ θα προκύψει η πλειοψηφία στην Επιτροπή μας, αλλά πρέπει να κερδίσουμε την όλη υπόθεση και στην Ολομέλεια. Και αν τελικά τα θέματα εδώ τα ε, ταλαιπωρούμε υπερβολικά, φοβάμαι ότι τελικά όταν πάνε στην Ολομέλεια καταπίπτουν. Ένα άλλο θέμα που θέλω επίσης ε, να θίξω και που έχει, υπάρχει πρόβλημα για μας είναι το θέμα των μεταβιβάσεων. Κατανοούμε βέβαια ότι εκεί όπου εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί, τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν μόνα τους κατά πόσον θα επιβάλλουν όρους ή όχι. Όμως η πρόταση που έχει κατατεθεί αφορά και εκείνα τα κράτη-μέλη ε, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερα να αποφασίσουν. Δηλαδή, αν θέλετε με άλλα λόγια, είναι ένα βήμα προς τα πίσω όσον αφορά στην κοινή αγορά. Και πρέπει να σεβόμεθα τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών Θεωρώ ότι τα ίδια τα κρατημέλη έχουν μια πολύ καλή γνώση τη αγορά εργασία στα ίδια και γι' αυτό ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Κατόπιν τούτου, τι συμβαστικές προτάσει που αφορούν στο θέμα αυτό θα τι απορρίψουμε. Κάτι άλλο που ετέθη, το θέμα της εκπαίδευση. Εμείς ως φιλελεύθεροι είμαστε πρόθυμοι να προχωρήσουμε περισσότερο, δηλαδή ε, να προβλέπεται δεσμευτικά η εκπαίδευση διάρκειας πέντε ημερών. Και αυτό δεσμευτικά, διότι πιστεύω ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, όπου η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση είναι καθοριστική σημασίας, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ακριβώς εδώ πρέπει να πούμε δεσμευτικά ότι θέλουμε να προσφέρουμε αυτή την εκπαίδευση εκπαίδευση στους εργαζομένους. Κατόπιν τούτου, η διατύπωση που επελέγει στην τροπολογία, η σχετική διατύπωση είναι αποδεκτή, αλλά εγώ θα προτιμούσα να προχωρήσουμε περισσότερο. Γιατί σε τελική ανάλυση, γιατί γίνεται αυτή η επανεξέταση. Υπάρχει διότι επιθυμούμε στις ε, υπηρεσίες εδάφους ε, να υπάρχει καλύτερη ποιότητα. Μέχρι τώρα ε, δεν ήταν ικανοποιητικό το επίπεδο της εκπαίδευσης. Δηλαδή μερικοί λένε εντάξει δύο μέρες φτάνουν και μετά να δούνε τέλο πάντων τα κρατημέλη τι μπορούν να προσφέρουν. Όμως είτε θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα είτε όχι. Αν το θέλουμε τότε θα πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των εργαζομένων. Εμείς ως φιλελεύθεροι θέλουμε να κάνουμε αυτό το βήμα, θα στηρίξουμε αυτή την τροπολογία. Θα θέλαμε βέβαια να είναι ακόμα πιο φιλόδοξη. Μερικές φορές έχουμε δύσκολους ε, συμβιβασμούς. Ο Τόμας Χέντελ. Όσον αφορά αυτά που είπε η προραλήσια σας, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, αν δούμε λιγάκι ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη προσφέρεται εκπαίδευση δύο ημερών και μόνο και έχοντας κατά νου ότι εδώ μιλάμε για έναν τομέα που είναι καθοριστικός για την ασφάλεια, καταλαβαίνετε ότι οι πέντε μέρες είναι το ελάχιστο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ε, συμφωνώ με την συνάδελφο Σπάι όσον αφορά το θέμα αυτό. Και επανέρχομαι στην αρχή. Θα ήθελα να επισημάνω τις συζητήσεις που κάναμε στις ακροάσεις και στην Επιτροπή μας. Εκεί δηλαδή που τοποθετηθήκαμε στην ουσία της οδηγίας. Και εκεί συμφωνήσαμε σχεδόν όλοι ότι υπάρχει μια σειρά θεμάτων τα οποία μπορούν να βελτιωθούν αυτή τη στιγμή. Γιατί η τελευταία απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον σε κάποια κράτη-μέλη, σε πολλούς ε, απασχολούμενους ε, στους αερολιμένες οδήγησε ε, στο να επιβληθεί dumping και το 40% των εργαζομένων, στη Γερμανία τουλάχιστον, ε, μπορούν να επιβιώσουν μόνο εφόσον λάβουν συμπληρωματικά κοινωνικά επιδόματα. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάθε λόγος σε αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις διατάξεις. Βέβαια, το θέμα που τίθεται είναι το εξής. Ε, πρέπει μήπως όλο αυτό το θέμα να το απορρίψουμε ή πρέπει να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Και τελικά καταλήξαμε στο να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την οδηγία. Νομίζω λοιπόν η ουσία της ε, βελτίωσης μπορεί να λάβει χώρα εδώ, στην Επιτροπή μας. Βεβαίω ε, σέβομαι πολύ και ιδιαίτερα αυτά που έχει προσφέρει ο κύριος Τόμας Μαν, τον κόπο του. Και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος με κάποιες ε, μορφές διατύπωσης και δεν καταλαβαίνω γιατί οι τομείς που μέχρι τώρα δεν ρυθμίζονται, γιατί αυτοί να μην πρέπει να συμπεριληφθούν μαζί με τους άλλους στην ε, πλήρη ρύθμιση και, στην, ε, και στον έλεγχο. Θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την απασχόληση και την κυρκή κατάσταση των εργαζομένων στους αερολιμένες. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή αυτή έχει ένα πραγματικά σημαντικό καθήκον. Ε, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει στην Επιτροπή Μεταφορών. Η δική μας θέση στην Ολομέλεια μπορεί να αλλάξει αν τελικά μετά από τις προτάσεις που θα μας ε, κατατεθούν ε, αλλάξει κάτι. Γιατί αν δεν αλλάξει τίποτα παραμένουμε στη θέση μας που είναι από το τίποτα καλύτερα έστω το κάτι. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέρ είναι εδώ. Από την Κομισιόν μπορεί να μας πει περίπου πόσο έχει η συζήτηση στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, πρώτο σημείο για το που βρίσκεται η συζήτηση σε επίπεδο Συμβουλίου. Το Συμβούλιο ενέκρινε μια γενική προσέγγιση κατά το Συμβούλιο Μεταφορών του Μαρτίου και γενικά ακολουθώντας την ίδια γραμμή με την Κομισιόν. Ένα άνοιγμα που να μην είναι ένα απόλυτο άνοιγμα των ε, αγορών, των δημοπρασιών, αλλά να έχουμε έναν δεύτερο προμηθευτή. Και το Συμβούλιο θέλει να εισάγουμε και μία διάταξη σχετικά με τις μεταφορές που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν ε, για τις ε, μεταθέσεις προσωπικού για τις ε, περιορισμένες υπηρεσίες. Επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι η θέση της Κομισιόν είναι μια ισορροπημένη θέση. Εμείς εδώ έχουμε μια πραγματικότητα σε πολλά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε λέξη που γράφεται ε, έχει επιπτώσει στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα αυτών των αεροδρομίων και η Κομισιόν επέμεινε να ξεκαθαρίσει όλες τις διατάξεις που αφορούν στις μεταφορές ούτως ώστε να μην υπάρχει επίπτωση του κοινωτικού δικαίου σε αυτόν τον τομέα. Βασιστήκαμε στην οδηγία του 96 για το θέμα της υπεργολαβίας, για την διάρκεια και τον σεβασμό των ε, συλλογικών συμβάσεων και για το θέμα της ποιότητας όπως και για το θέμα της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών εδάφους ε, που να είναι υπηρεσίες ε, καλές για τον επιβάτη. Πρόκειται για μία πολύπλοκη νομοθεσία για το θέμα της κατάρτισης μας λέτε να προχωρήσουμε περισσότερο. Εμείς έχουμε εισάγει δύο σημεία στην κατάρτιση σχετικά σχετικά με την έγκριση Πρέπει λοιπόν εμείς στη διαδικασία της συναπόφασης να τονίσουμε αυτήν την... να εγκρίνουμε σε συναπόφαση αυτή την νομοθεσία. Το κοινοτικό δίκαιο δεν πρέπει να εμποδίζει αφενός τις μεταθέσεις, αλλά δεν πρέπει να τις επιβάλλει. Μόνο ένα κράτος μέλος τάχθηκε υπέρ των υποχρεωτικών μεταθέσεων σε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι διατάξεις ε, που είναι συνδεδεμένες με το άρθρο 40 είναι διατάξεις ιδιαίτερα παροχημένες και παρισφρίουν στην ε, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα των κρατών μελών. Το να αποφασίζει κανείς να απαγορεύει τις απολύσεις στις υπηρεσίες εδάφους για λειτουργικά θέματα ξεπερνάει τα όρια της οδηγίας 2023. Αν θέλετε να ενισχύσουμε τον τομέα της κατάρτισης, έχουμε ένα μεγάλο περιθώριο για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους. Τώρα για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι δύσκολο και συνδυάζεται και πολύ δύσκολα με τις θέσεις που έχει μέχρι τώρα λάβει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε ότι είναι ένα, πολύ, ένα πολύπλοκο θέμα. Να δούμε πώς θα, περάσει, πώς θα γίνει η διαπραγμάτευση όταν εγκρίνουμε εμείς τη θέση μας. Εμείς θα ψηφίσουμε αύριο. και στη συνέχεια η Επιτροπή Μεταφορών θα αποφασίσει στις 8 Οκτωβρίου. Κύριε Τόμας Μαν, δεν σας ξανάδωσα το λόγο. Συγγνώμη. Επιτρέψτε μου σύντομα να πω κάτι. Κοιτάξτε, αυτή είναι η μοίρα των ε, συμβιβασμών. Στο Κοινοβούλιο ε, μας κατηγορούν ε, οι δημοσιογράφοι ότι είμαστε απέσιοι. Ε, Κοιτάξτε, οι συμβασμοί αυτοί δεν έχουν προκύψει με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά ε, προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μια κοινή γραμμή. Βεβαίως ε, και υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Νάντια, εσείς οι φιλελεύθεροι θελήσατε να πείτε ότι οι δύο ημέρες φτάνουν. Εμείς είπαμε πέντε και συμφωνήστε. Ήδη αυτό είναι ένα βήμα προς τα πάνω αν είχαν συμφωνήσει οι υπόλοιποι στην δική σου ομάδα με αυτό που είπες, τότε από τις πέντε θα είχαμε πάει ακόμα πιο πάνω. Ακόμα και στη δική μας την πολιτική ομάδα δεν συμφωνούμε όλοι και αυτό είναι σαφές. Άρα δηλαδή νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά. Εγώ απλά επιθυμώ μια πολιτική ομάδα που λέει ότι δεν επιθυμούμε να υπάρχει πρόταση κανονισμού της Επιτροπής. Ε, αγαπητή Τζίνς, ε, θα ήθελα να το ξαναδείς λιγάκι. Γιατί σε μια συμβαστική πρόταση αυτό που παίζει ρόλο είναι να γίνει ένα βήμα και να υπερψηφιστεί η πρόταση. Και έκαναν και κάποιου ε, υπολογισμού, Δηλαδή, αν συμφωνήσουν οι πολιτικές ομάδες, έστω και αυτέ που είπαν ότι θα ψηφίσουν με το ζόρι, ε, αυτό δεν μετράει, το αποτέλεσμα μετράει, εκ του αποτελέσματο κρίνονται. Ε, γιατί άλλο να πει κανεί ναι και άλλο όχι ή απέχω. Σε τελική ανάλυση, επειδή χρειαζόμαστε πάρα πολλού, σα είπα, έκανα του υπολογισμού μου και εάν τελικά ε, δεν αλλάξετε θέση, θα βρεθεί άλλη επιτροπή που θα είναι αρμόδια και όχι δικιά μα. Ε, αυτά που βρίσκω πολύ σημαντικά είναι οι συλλογικέ ε, προτάσει. Ε, είπαμε ότι στου αρολιμένε υπάρχουν διαφορέ και δεν θέλουμε την ασύντοτη απελευθέρωση, αυτό που επιθυμούν άλλοι. Όχι αυτό. Τα χαιρόμουν λοιπόν πάρα πολύ αν μπορούσαμε να πούμε ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν εμείς τελικά καταλήξαμε έτσι ώστε να μην υπάρξει εφήμωση να μπορούμε να πούμε ότι πράγματι ε, ο κύριος Μαν έχει δίκιο και μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους ότι εμείς ε, θα δουλέψουμε έτσι ώστε να έχετε δίκαιες απολαβές και να μπορούμε να ε, διαβεβαιώσουμε και τους επιβάτες ότι στους αερολιμένες θα έχουν ικανοποιητική ποιότητα. Αν το κατορθώσουμε αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Ίσως σήμερα το βράδυ να γίνουν κάποια σχετικά τηλεφωνήματα. Ελπίζω γιατί θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα και ελπίζω στην Ολομέλεια να έχουμε μεγαλύτερη συνένεση από αυτό που φαντάζονται μερικοί. Εάν κατάλαβα καλά, θα περάσετε μια ιδιαίτερα δυναμική νύχτα. Και έχουμε λοιπόν σας μέχρι αύριο για την ψηφοφορία. Πάμε στο σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη η συνάδελφος Μπίργκιτ Σίπελ θα μας παρουσιάσει τις τροπολογίες, συμβιβαστικές τροπολογίες, για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Έχετε το λόγο, συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να πω το εξής. Όσον αφορά στις ε, διαπραγματεύσεις, οι διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή είχαμε μεγάλη πίεση και ε, όλο το Σαββατοκύριακο δουλεύαμε πάνω στους, ε, στις προτάσει. προτάσεις και διαπιστώσαμε ότι για πάρα πολλά θέματα όχι μόνο είχαμε διαφορετική θέση αλλά εν μέρη και ε, αντίθετες απόψεις, εκ διαμέτρου αντίθετες. Ακριβώς λοιπόν επειδή το θέμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ακριβώ επειδή υπήρχαν εκδιαμέτρου διαμέτρου αντίθετες απόψεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες ε, και τους ε, συνεργάτες για τη συνεργασία, γιατί με την συνεργασία αυτή και με την ανταλλαγή των email κατορθώσαμε να έχουμε μπροστά μας 24 συμβαστικές ε, τροπολογίες που αποτελούν πραγματικά συμβασμό. Μερικοί λένε ότι είναι πάρα πολύ προχωρημένες, άλλοι πάλι όχι, αλλά ο κύριος Μαν είπε και ο ίδιος ότι αυτό σημαίνει συμβασμός. Αυτό που κατορθώσαμε, και νομίζω αυτό είναι καλό για την Επιτροπή, κατορθώσαμε σε αυτή την ε, ανάθεση δημόσιων συμβάσεων να αναφέρονται τα κοινωνικά κριτήρια. Όχι πάντα δεσμευτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρονται και στις αιτιολογικές σκέψεις, εξηγούνται ακριβώς τι είναι αυτά τα κοινωνικά κριτήρια. Νομίζω λοιπόν ότι στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται μόνο ε, τα περιβαλλοντικά κριτήρια και καθόλου τα κοινωνικά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τουλάχιστον σε κάποια σημεία αναφέρονται τα κοινωνικά κριτήρια. Εκτός αυτού η πλειοψηφία συμφώνησε ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η κατατόπουση ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και οι, λογικές, και οι συλλογικές συμβάσεις. Αυτό είναι ένα καλό βήμα. Οφείλουμε να το αναφέρουμε ως Επιτροπή Απασχόλησης. Και όσον αφορά ε, την αιτιολόγηση κατακύρωσης ε, του διαγωνισμού ή αποκλεισμού, στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κρίνεται άγωνος, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρονται ε, και άλλα κριτήρια, όπως παραδείγματο χάρη το ότι υπάρχει κίνδυνος να μην καταβάλλονται οι αποδοχές των εργαζομένων. Ε, αυτός ο λόγος είναι λόγος αποκλεισμού, μόνο βέβαια εφόσον η επιχείρηση ε, καταδικάζεται τελεσίδικα. Υπάρχει η σύμβαση του ε, Διεθνού Γραφείου Εργασία η 94, 94, την οποία όμω δεν έχουν υπογράψει όλα τα κράτη-μέλη. Και εμείς ε, περιλαμβάνουμε μια παραπομπή σε αυτήν την ε, σύμβαση. Κανείς δεν εμποδίζεται να την εφαρμόσει και αν το κάνει αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα βελτίωσης. Εξάλλου συμφωνήσαμε η αρχή του μειοδότη να διαγραφεί από το κείμενο, να μην ισχύει ε, η κατακύρωση στο μειοδότη. Αυτό που δεν κατορθώσαμε ήταν στο θέμα της μείωσης των ε, υπεργολάβων και στην ε, ανάληψη ευθυνών από πλευράς υπεργολάβων. Νομίζω ότι με τη συμβαστική πρόταση αυτή έχουμε τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα που είναι πολύ καλύτερο από το ισχύον κείμενο για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Και νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα όταν θα ολοκληρωθούν οι κατάλογοι ψηφοφορίες αύριο θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν θα χοροπηδήσουμε από τη χαρά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε στα χέρια μας κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή Καλό λοιπόν, θετικό το αποτέλεσμα. Η Νάντια Χίρς, από ο σκιώδης των φιλελευθέρων, ή μάλλον εξ ονόματος του σκιώδου, συζητητή από των φιλελευθέρων, θα ήθελα να πω τα εξή. Έχουμε λάβει τα σχέδια συμβαστικών τροπολογιών και έχουμε καταλήξει τα εξή συμπεράσματα. Πρώτον, υπάρχουν 12 συμβαστικές που μπορούμε να υποστηρίξουμε ως ομάδα η CGAGA λέει VWX and on... και αντίθετα τις εξής τροπολογίες ε, E, um, because it does not... Ε, Όπω η B παραδείγματο χάρη δεν μπορούμε να τι υποστηρίξουμε διότι η συγκεκριμένη δεν λαμβάνει υπόψη την τροπολογία 11 τη Μαρία Χάρκιν, την τροπολογία C δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε γιατί παραπέμπει στη σύμβαση τη Διεθνού Οργάνωση εργασία και των σχετικών διατάξεων για την απασχόληση που είναι εφαρμοστέ στο κράτο μέλο, όπου ε, διεξάγονται τα έργα τη σύμβαση. και αυτέ οι δύο μνήε δημιουργούν νομική ανασφάλεια σε σχέση με την οδηγία για την απόσπαση. FHM και U τώρα. Αυτέ οι τροπολογίε επίση δεν μπορούν να υποστηριχθούν για τον ίδιο λόγο, επειδή παραπέμπουν σε διατάξει για την απασχόληση που ισχύουν στο κράτο μέλο όπου θα διεξαχθούν τα έργα ή που θα παρασκευθούν οι υπηρεσίε και έτσι δημιουργείται νομική ανασφάλεια. Στη συνέχεια, τροπολογία ε, Α δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε, διότι καταργεί το κριτήριο του χαμηλότερου κόστου ε, και εισαγάγει νέα κοινωνικά κριτήρια. Η ΕΜΕ Επίση, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ούτε και η ΖΗ, διότι οι υπεργολαβίε δεν μπορούν να γίνουν δεκτέ. δεν μπορούμε να προδικάσουμε την έκβαση των συζητήσεων για την ε, σχετική οδηγία. Συμβαστική τροπολογία πει δεν είναι αποδεκτή, διότι αναφέρεται ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίσουν ε, την ε, συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσει. Εμεί σε ορισμένες περιπτώσεις θα θέλαμε ισότητα ανάμεσα σε όσοι υποβάλλουν προσφορές ε, και τι δύο συμβαστικέ τροπολογίες ε και ε, ε, ζ. μάλλον παραπέμπουν στην αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν συνάδουν με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων και αν γίνουν οι διαγραφές όπως προτείνεται σε αυτές τις δύο τροπολογίες δημιουργείται ακόμη περισσότερη νομική ανασφάλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Madam and thank you to... Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε την Πύρκη Τσίπελ, την εισηγήτριά μας. Ε, εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο και όπως είπε ήδη, ε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Ε, το ΕΛΚΑ μπορεί να υποστηρίξει ή μάλλον, όσε οι τροπολογίε υποστηρίζονται από το ΕΛΚ μα βρίσκουν και εμά σύμφωνος. Όπως είπε η κυρία Σίπελ, θέλω να τονίσω τη σημασία της συμβαστική ΣΥ που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό αυτέ αυτές οι αρχές για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων να εκφράζονται με ενάργεια, όπως ε, στη φρεσολογία τη συμβαστική. Ε, θα θέλαμε να ε, έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων σε σχέση με την διατύπωση που σχετίζεται με τη Σύμβαση Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ε, στην επόμενη τροπολογία. Είμαι ε, σχεδόν σίγουρη θα μπορούσε το Συμβούλιο να δεχθεί την ε, τροπολογία μας. Τροπολογία τώρα 1. Έχουμε τους υπεργολάβους, τη ρήτρα για τις υπεργολαβείς και το σχετικό άρθρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο βασικός εργολάβος να παράσχει ε, τις πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους, ε, δηλαδή τα ονόματά τους, ε, τα στοιχεία τους, το νόμιμο εκπρόσωπό τους, ε, διότι το άρθρο περί υπεργολαβίας είναι πλέον τόσο ξεκάθαρα διατυπωμένο και αυτό ήταν και ο, αυτός είναι ο λόγος ε, που δεν υποστηρίζαμε εμείς ε, στα περί κοινής ευθύνης, ε, διότι υπερβαίναμε την κείμενη νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Τώρα όμως που ρυθμίστηκε το θέμα και είμαι σίγουρη ότι με αυτό το άρθρο θα διαλευκανθεί η υπόθεση και ελπίζω στην ΙΜΚΟ να γίνει δεκτή αυτή η συμβαστική τροπολογία. Θέλω επίσης να αναφερθώ στην αλφα παρότι αναφέρεται στα εκτιμώντας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε τα διάφορα κριτήρια όπως ε, τα κοινωνικοπεριβαλλοντικά κριτήρια. Να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή ότι αν οι αναθέτουσες αρχές επικαλούνται αυτά τα κριτήρια, θα πρέπει να γίνει με τρόπο σαφή για όλους. Στους διαγωνισμούς όπου θα υπο... ούτως ώστε αυτοί που υποβάλλουν προσφορές για διαγωνισμούς να γνωρίζουν ακριβώ τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν για την επιλογή. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι στο κατάλογο ψηφοφοριών έχουμε μια σειρά τροπολογιών, όμως ακούσαμε ήδη ότι διάφορες ε, τέτοιες τροπολογίες δεν ε, εμπίπτουν καν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Ε, οπότε είτε θα αποσυρθούν είτε θα κρυθούν μη παραδεκτές ευελπιστώ ότι στην αυριανή ψηφοφορία θα είναι συντομότερο ε, ο κατάλογος ψηφοφοριών ε, σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα. Ε, Μπίργκετ και πάλι συγχαρητήρια, ήταν δύσκολο το έργο σου, αλλά τα κατάφερε σε εξαίσια. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, μιλήσατε όλοι. Ξαναδίνω το λόγο στην εισηγήτρια. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής, ότι για μένα είναι σημαντικό να αναφερθώ σε δύο θέματα. Η συνάδελφος από τους οι συνάδελφοι γενικότερα, είπαν ότι θα προκύψει νομική ανασφάλεια αν γίνεται αναφορά στις κατατόπους ισχύουσες ε, διατάξεις. Κοιτάξτε, ε, υπάρχουν όμως και άλλα άρθρα όπου αναφέρεται, όπου εργοδότης ε, είναι υποχρεωμένος ε, στους ε, μετέχοντες ε, να τους ενημερώσει για τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, κυρίως περιεργασίες, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων. Και από πλευράς Γερμανίας θέλω να σας πω ότι πολύ συχνά προκύπτει στρέβλωση ανταγωνισμού λόγω του ότι δεν τηρούνται οι επιτόπου ισχύουσες λογικές συμβάσεις και οι προϋποθέσεις. Γιατί πολύ συχνά αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού γιατί είναι πάρα πολύ ακριβές. Κατόπιν τούτου υπάρχει το θέμα του ανταγωνισμού που όπως σας είπα μπορεί να το δει κανεί από δύο διαφορετικές ε, πλευρές. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τους ε, κοινωνικούς φορείς, νομίζω ότι το όλο αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Εμάς ως ε, ε, Κοινωνική Επιτροπή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα γιατί αυτό που παίζει ρόλο είναι να υπάρχει απασχόληση για άτομα με αναπηρία ή με άλλου είδους προβλήματα τα οποία προσωρινά τουλάχιστον δεν έχουν ε, καμία ευκαιρία να εργαστούν. Ε, και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικές αυτές οι διατάξεις που αναφέρονται στην αποφυγή της ε, στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και είμαι πραγματικά περίεργη να δω πόσο μακροσκελής θα είναι αύριο ο κατάλογος ψηφοφορίας. Καλό κουράγιο για όσους φτιάξουν αυτόν τον κατάλογο ε, ψηφοφορίας. Η αρμόδια επί της ουσίας ΙΜΚΟ θα ψηφίσει 10 Οκτωβρίου, εμείς αύριο. Πάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να συζητήσουμε για 5 συμβιβαστικές τροπολογίες επί 133. Πρόκειται για την έκθεση της συναδέλφου Μανέσκου για τις ε, συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς ε, του ύδατος της ενέργειας των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η Νάντια την καθιστά την κυρία Μανέσκου, η οποία δεν μπορεί να είναι παρούσα. Ευχαριστώ. Από εξ ονόματο τη εισηγήτριά μα, τη κυρία Μανέσκο, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω του σκιώδει εισηγητέ ε, για την καλή συνεργασία που είχαν. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερι συμβαστικέ τροπολογίε ε, ε, το ΕΛΚΑ και οι σοσιαλιστές έχουν υποστηρίξει το περιεχόμενο. Ο στόχος ήταν να συμπεριλάβουμε συμβαστικές τροπολογίες ε, και τις τροπολογίες ε, που θεωρούμε ότι είναι πρόσφορες και συνδέονται άμεσα με το έργο της Επιτροπής μας. Συμβαστικές τροπολογίες, άρα μας ενδιαφέρουν διότι αναφέρονται στο εκτιμώντας 4, όπου τονίζεται ο ρόλος των δημοσίων συμβάσεων, το άρθρο 1 σε σχέση με τις συμβάσεις που σχετίζονται με τις εταιρείε κοινωνικού περιεχομένου, άρθρο 5 παράγραφος 1 για τις εταιρείε για την ετικετοθεσία, 13.1 ε, για την επιλογή των συμμετεχόντων και την σύνταξη των ε, συμβάσεων και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε ε, για αυτήν την έκθεση. Θα ήθελε κάποιος το λόγο, παρακαλώ. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is a nevében szólok, aki éppen Θα ήθελα να εκπροσωπήσω τον ασκιώδη συγκητή μα, ε, διότι ψηφίζει αυτή τη στιγμή σε μια άλλη επιτροπή και δεν μπορεί να παρευθεί στη συζήτηση. Όπω είπε και η κυρία Χίρ, ήταν πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στην εισηγήτρια και του σκιώδη εισηγητέ. Το ΕΛΚ υποστηρίζει και τι τέσσερι τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Φρανσουάς Καστέξ. Υποστηρίζουμε επίσης το συμβιβασμό. Υπήρξε ένα καλό κλίμα, είχαμε μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Λυπούμεθα όμως που οι αναφορές στο πρωτόκολλο 26 και στο ΙΣΕΖ δεν συμπεριλήφθηκαν επαρκώς στον συμβιβασμό. Θα ψηφίσουμε και άλλες τροπολογίες οι οποίες είναι σαφέστερες και δεν συμπεριλήφθησαν στον συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ουχή. Η κυρία Χίρς δεν έχει τίποτα να προσθέσει. Ελπίζω η κυρία Μανέσκου θα ενημερωθεί για την ανταλλαγή απόψεων και ψηφίζουμε αύριο με το ίδιο χρόνο διάγραμμα της έκθεσης Σίβελ. Ο κύριος Μπέκερ ήρθε. Πάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. όπου συζητούμε την έκθεση Μπέκερ, πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την πρόθεση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ που δείξατε κατανόηση να αναβάλλετε λίγο τη δική μου την ομιλία, γιατί ξέρετε εγώ δεν έβρισκα καλύτερη πτήση για να φτάσω νωρίτερα. Τώρα, όσον αφορά τον τίτλο της δικής μου της έκθεσης, ε, αυτό που παίζει ρόλο και αναφέρεται είναι να υπάρχει καλύτερο κλίμα για τις ε, κοινωνικές επιχειρήσεις. Θέλω να επενέσω την Κομισιόν που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και θέλω επίσης να επισημάνω ότι με τις 283 τροπολογίες και με τους 29 συμβιβασμούς από όλες τις πολιτικές ομάδες ε, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα ε, και στο σημείο αυτό επιτρέψουμε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ε, και τις σκιώδεις εισηγήτες. Να ευχαριστώ θερμά τη γραμματεία του ΕΛΚ γιατί έκανα μια πάρα πολύ καλή εμπειρία εφόσον αυτή είναι και η πρώτη μου έκθεση. Κοινωνικές λοιπόν επιχειρήσεις. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ε, χαρακτηρίζονται από ένα ανεξάντλητο δυναμικό κυρίως ε, στον τομέα της ε, πράσινης και της άσπρης αποκαλούμενης οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας για τους νέους. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με τον ορισμό των κοινωνικών επιχειρήσεων. θελήσαμε να κάνουμε τον συντονισμό με άλλες ρυθμίσεις του παρελθόντος ε, και προσπαθήσαμε όλα αυτά να τα ε, εντάξουμε σε ένα και μόνο πλαίσιο. Ε, θα ήθελα να φερθώ σε μερικά σημαντικά θέματα, τα οποία προχωρούν και πέρα από την απλή προσφορά θέσεων εργασίας. Ρόλο λοιπόν θα παίξει η καινοτομία. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν καινοτομία. Και όλοι όσοι ασχοληθήκαμε με την έκθεση θέλουμε να επενδύσουμε στην καινοτομία γιατί πιστεύουμε ότι αυτές οι εννέα προϋποθέσεις τόσο αυτής της έκθεσης αλλά και άλλων του εκθέσεις που αφορούν στο Ταμείο Επενδύσεων και πολλά άλλα όλα αυτά θα προσφέρουν τη δυνατότητα να υπάρξουν νέες εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν σε θέματα ε, εργαζομένων, επανεπένδυσης, ε, προσφοράς, σε όλα αυτά έχουμε σαφείς και ανοιχτές ρυθμίσεις οι οποίες κρίνονται κυρίως από το ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να αποκαλείται κοινωνική εάν δεν μπορεί να αποδείξει ότι προσφέρει ότι έχει κοινωνική προσφορά. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με δυνατότητες ε, χρηματοδότησης, τις προτάξαμε αυτές, τις προβάλαμε, ε, ασχοληθήκαμε με την ε, θεμελιώδη έρευνα και τελειώνοντας θέλω να πω αυτό που παίζει ρόλο κυρίως είναι η επικοινωνία. Ε, πλατφόρμες ε, βέλτιστων ε, πρακτικών, συγκέντρωση δεδομένων και πολλά άλλα μέτρα τα οποία αφορούν τους πολίτες. Νομίζω ότι τελικά, λόγω του ότι τόσο τώρα όσο και στο μέλλον θα υπάρξει ανάγκη για κοινωνικά προϊόντα, νομίζω λοιπόν με αυτήν την έκθεση δημιουργούμε πλέον νέες προϋποθέσεις και θα κατορθώσουμε πάρα πολύ εύκολα οι νέοι στο μέλλον να ασχολούνται με, ε, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό απλά και μόνο διότι θα έχουν δημιουργηθεί και οι σωστές προϋποθέσεις. Ελπίζω ότι και νέοι μπορούν να ξεκινούν τέτοιου είδους περιπέτειες χωρίς ιδιαίτερη υποστήριξη η Κίνγκα Κούντς και μετά η Νάντια Χίρς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέκερ, τον εισηγητή μας, γιατί έδειξε πολύ ανοιχτό πνεύμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όπως σωστά είπατε, ήταν υψηλότατος ο ρυθμός των τροπολογιών που υπέβαλαν οι πολιτικές ομάδες. Ε, τώρα έχουμε περιοριστεί σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Ε, ελπίζω να τύχουν ευρύτητα της υποστήριξης. Έχουμε πλέον και έναν ορισμό ε, που ευθυγραμμίζεται με τον ορισμό για την κοινωνική καινοτομία. Ο ορισμός λοιπόν των κοινωνικών επιχειρήσεων και ορισμός για την κοινωνική καινοτομία αλληλοσυμπληρώνονται. Επίσης, απηχούνται πλέον οι προτεραιότητές μας, δηλαδή αφενός ε, θα ήταν σημαντικό να σχηματίσουμε μια πλήρη εικόνα του γενικότερου τοπίου και των προκλήσεων του τομέα αυτού. Δεν έχουμε αρκετούς νέους, παραδείγματος χάρη, να μια μεγάλη πρόκληση, οπότε δεν είναι αρκετά ελκυστικός ο τομέας για αυτούς τους νέους. Καλό θα ήταν να είχαμε και ένα είδος οικονομικής σταθερότητας ε, στον τομέα. Και τώρα εμείς εξετάζουμε ε, το θέμα για να συνειδητοποιήσουμε με ποιο τρόπο θα έπρεπε να κινηθούμε για να καλύψουμε και ομάδες, ε, κοινωνικές ομάδες όπως αυτή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αλλά σημαντικά ζητήματα είναι αυτό του κοινωνικού διαλόγου, παραδείγματο χάρη τη επαγγελματική ε, κατάρτιση, ε, τη επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών ε, δεξιοτήτων όλων όσων απασχολούνται σε αυτό το τομέα. Μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις και την πολύ καλή προετοιμασία είμαι πολύ αισιόδοξη για την έκβαση της αυριανής ψηφοφορίας. Πρόεδρος. Α, να, ε, αλλάζουμε λίγο το στυλ σε σχέση με ε, προηγούμενες ε, συζητήσεις εφόσον είστε αισιόδοξοι. Κύριε Χέρς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο κύριο Μπέκερ για την καλή συνεργασία οι συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και δύσκολες μάλιστα κυρίως για τους διερμηνείς και πιστεύω ότι αυτό αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του όλου θέματος. Και είναι πολύ καλό το ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχοληθήκαμε σε βάθος με αυτό το θέμα και με τις ε, διάφορες έννοιες, τους ορισμούς, γιατί καταλήξαμε τελικά ακόμα και σε φιλοσοφικές ε, συζητήσεις, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι οι πολίτες όλο και περισσότερο απαιτούν τέτοιου είδου ορισμούς όσον αφορά ε, στην κοινωνική επιχείρηση. Η έκθεση λοιπόν αποτελεί μια πολύ καλή πρωτοβουλία ε, και χαίρομαι που εμείς ως φιλελεύθεροι μπορούμε να υπερψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες. Η συνάδελφος η προλαλήσασα ανέφερε πολλά σημαντικά πράγματα. Εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε μια κατεύθυνση ε, που πάρα πολύ εκτός κοινοβουλίου ε, την βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρουσα. Στο μέλλον λοιπόν ίσως όλοι συνειδητοποιήσουν ότι αυτός είναι ο μόνος ένας και παρτός δρόμος. Άλλοι θέλουν το λόγο. Όχι. Κύριε Σιγητά, θέλετε να πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, και για τις ε, προτάσεις που καταθέσατε ακόμα και σήμερα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι κατέθεσαν τις απόψεις τους. Εμείς προφανώς όλα αυτά θα τα λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη συνεργασία και παρακαλώ την ε, Επιτροπή να δώσει την ευρύτερη δυνατή συνένεσή της, γιατί αυτό θα αποτελεί μήνυμα προς τα έξω το πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ κύριε <coughs> Θα ψηφίσουμε αύριο. Σε ένα πλαίσιο διότι εμείς ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την σχετική έκθεση που συνδέεται με αυτό το κείμενο και μετά συμβατά αυτά με την ε, διαδικασία που μας ε, πρότεινε ο Επίτροπος και που καλύπτεται από άλλες εισηγήσεις, από άλλες εκθέσεις, Σε αυτό το πλαίσιο ελπίζουμε ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξατε σε συνεργασία με τις άλλες ομάδες να εμπνεύσει το κείμενο του Επιτρόπου και θα δούμε πώς αντιδρούμε σε αυτήν τη νέα θέση, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης και έχουμε εδώ τις συνδυαστικές τροπολογίες για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Επαναλαμβάνει τον τίτλο στα γαλλικά η Πρόεδρος και δίνω το λόγο στην Κίνγκα Γκόντς. Σας ευχαριστώ. Θα κάνω μόνο μία σύντομη περίληψη για το πρόγραμμα, για το οποίο γνωμοδοτούμε με αποδέκτη την Επιτροπή Πολιτισμού. Είναι μεγάλη επιτυχία το Media και ε, Media Mundos. Αυτά τα δύο προγράμματα ε, έτυχαν μεγάλες υποστήριξεις και ε, το σχέδιό μας επικεντρώνεται γύρω από την ε, ιδέα της δημιουργικής βιομηχανίας, να γίνει πιο ανταγωνιστική δηλαδή και να απασχολεί περισσότερους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της κρίσης για να προαγάγουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργία μας και να προσανατολιζόμαστε προς την ανταγωνιστικότητα. Είχαμε μακροσκελέστατη συζητήσουμε με τους και τους για αυτό το θέμα. Ε, είναι μεγάλο το δυναμικό της δημιουργικής αυτής βιομηχανίας και συμφωνήσαμε ω επιτοπλιστών σχετικά με το ότι μέσω καταρτήσεων ή ε, μέσω κάποιας ε, μορφής αρρωγής θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου αυτού. Νομίζω ότι μετά από τις συζητήσεις ε, συμφωνήσαμε για το εξής, ότι εφόσον ε, μεταξύ άλλων ο βασικός μας στόχος είναι να μιλήσουμε για το θέμα της ανταγωνιστικότητας και να ε, βρούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμβάλλουμε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Κρίναμε λοιπόν ότι μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε από αυτόν, ναι, εκτός από τους ε, πρασίνους ε, και την ε, ΓΚΟΕ που δεν μπόρεσαν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Έχουμε την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων εκτός από αυτές τις δύο για, για άλλες συμβαστικές τροπολογίες. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη, οι τροπολογίες που σχετίζονται με την, το ρόλο των νέων παραδείγματο χάρη, ε, ή ε, το να ληφθούν υπόψη ε, ανα, ειδικέ ανάγκες σε κάποιων ατόμων. Επίσης, για τις τροπολογίες που σχετίζονται με τους νέους τρόπους παραγωγής αλλά και διανομής των έργων σε σχέση με τα επιχειρηματικά προσόντα, όλοι συμφωνούμε ότι έχουν καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής αυτονομίας ε, του κλάδου. Αυτά είναι όλα σημεία κλειδιά. Έχουμε, αυτή είναι, ε, αυτό είναι συνοπτικά το σχέδιό μας. Έχουμε 38 συμβαστικές τροπολογίες. Δύο μόνο δεν, μπορέ, δεν μπόρεσαν να τύχουν τις υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων. Όπως σας είπα διαφώνησαν οι πράσινοι και οι γκουε. Ναι, νομίζω και ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμο το έγγραφό μας και κυρίως για την Επιτροπή Πολιτισμού και κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου για τις τόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε για την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χίρσε είναι η μέρα σου σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και επίση και την εισηγήτρια για τη συνεργασία που είχαμε. Νομίζω ότι ε, συμπληρωθήκαμε πάρα πολύ καλά. Εμείς ε, ως ε, φιλελεύθεροι συμφωνούμε με τις συμβαστικές προτάσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτές. Για μας βέβαια υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα. Το στοιχείο του ανταγωνισμού και νομίζω αυτό είναι πολύ καλό για την παραγωγική επικοδομητική Ευρώπη. Είναι σημαντικό να υπάρχει το στοιχείο του ανταγωνισμού και από την άλλη βέβαια ε, να συμπεριλαμβάνονται οι νέοι σε προγράμματα ανταλλαγής. Ε, να γίνεται δηλαδή αυτό το βήμα προς τα εμπρός. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Ο κύριος Μπέκερ. Σας ευχαριστώ πολύ ε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί πράγματι και εδώ είχαμε πολύ επικοδηματικό ε, κλίμα συνεργασία και πολλές ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε συζητήσει. Υπάρχει το στοιχείο του ανταγωνισμού, ε, το οποίο χαρακτήρισε τις ε, μας. μα. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Το ένα είναι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η δημιουργική οικονομία πρέπει να προβάλλει τον ανταγωνισμό απέναντι και σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες εμπορικές δυνάμεις. Αυτό το ξέρουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κίνα, την Ινδία και από άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτό όμως δεν πρέπει να το κατανοούμε μόνο, αλλά και εμπορικά. Και βεβαίως ε, ο ανταγωνισμός πρέπει να αντιμετωπίσει και κάτω από το πρίσμα ότι υπάρχει μια κοινωνική υποχρέωση ε, την ε, οποία δεν βρίσκουμε μόνο ε, σε μια δημιουργική οικονομία. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε, όπως σας είπα, τον εξάντλητο δυναμικό και αυτής της οικονομίας. Ας πούμε, ε, στην Γερμανία η παραγωγική οικονομία έχει άμεση σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία που είναι και η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Ε, γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά παρακαλώ να τα έχουμε κατά νου όταν εξετάζουμε αυτή την έκθεση. Θα ήθελε κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Θα ψηφίσουμε αύριο ελπίζοντας ότι θα λάβει υπόψη της στις 9 Οκτωβρίου Επιτροπή Πολιτισμού. Κίνγκα θα ξαναήθελε στο λόγο. Όχι, δεν έχω άλλα σχόλια. Ευχαριστώ. Σημείο 8. Οπότε τώρα εγώ θα σας παρουσιάσω τις 8 συμβιβαστικές τροπολογίες ε, που συντάξαμε με τον Σκεώδη τι πρόκειται για τη δική μου γνωμοδότηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Πριν σας παρουσιάσω τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Να σας πω ότι για την Επιτροπή μας αυτή η γνωμοδότηση αποτελεί μία σημαντική συνεισφορά στην θέση του Κοινοβουλίου στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων. Δεν το λέω αυτό επειδή είμαι εγώ η εισηγήτρια. Η αποέλλειψη ταπεινοφροσύνη σας, σας το λέω γιατί εμείς επιλέξαμε να ακολουθήσουμε μία στρατηγική που μας οδηγεί να διαφοροποιήσουμε την διαπραγμάτευση για την νομοθετική βάση από τη διαπραγμάτευση του συνόλου του πακέτου για την πολιτική βάση. Για την νομοθετική βάση έχουμε μία ιδιαίτερα δυναμική ομάδα, κυρία Στάιλρουπ, κύριος Κώστα, κύριο, Άρκιν, κυρία Άρκιν, κύριε Σαρτιέ, Και εδώ πρόκειται για την εξέταση των βάσεων εκείνων τις οποίες είμαστε στη συναπόφαση με το Συμβούλιο και ξέρετε τις δυσκολίες μας να καταλήξουμε επί του συγκεκριμένου. Υπάρχει και η δική μας συνεισφορά σχετικά με τις διαπραγματεύσεις Κοινοβούλιο Κομισιόν και αφορά στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και, την και σε αυτήν τη φάση των διαπραγματεύσεων δεν θα σας διέφυγε ο Χέρμαν Βάρον Πόη συγκάλεσε στις 23-24 ε, Νοεμβρίου ένα έκτακτο συμβούλιο και υποχρέωσε την Κυπριακή Προεδρία να διορθώσει ε, μερικά πράγματα για το χρονοδιάγραμμα. Εμείς, από την άλλη μεριά όμως, και εμάς το Κοινοβούλιο μας αναγκάζει να πούμε ορισμένα πράγματα και να στείλουμε σαφή μηνύματα πριν από αυτήν την ε, προθεσμία 22-23 Νοεμβρίου. και υπό την ευθύνη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέσα στα πλαίσια της ομάδας επαφής που όπως ε, ξέρετε αποτελείται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους εισηγητές, τον πρόεδρο των προϋπολογισμών και σκεώδης εισηγητές ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμών αλλά και οι υπευθύνων των λεγόμενων τεχνικών επιτροπών. Συμφωνήθηκε λοιπόν σε την επιτροπή, ομάδα επαφής, να συντάξει το Κοινοβούλιο μία ενδιάμεση έκθεση που δεν θα αποτελεί την τελική μας θέση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά θα επιτρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα πριν από το Συμβούλιο της 22ης και 23 η Νοεμβρίου. Οι πολιτικές ομάδες θα κινητοποιηθούν για το περιεχόμενο αυτής της προσωρινής έκθεσης, που θα ψηφίσουμε τον Νοέμβριο στο Στρασβούργο, 16 ή 17 Νοεμβρίου πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά ως Τεχνική Επιτροπή φαίνεται ότι η ψηφοφορία μας αύριο θα αποτελεί και τη συνεισφορά μας σε αυτήν την ενδιάμεση έκθεση και αυτή είναι και η σημασία των βασικών μήνυμάτων που, που επιλέγουμε να στείλουμε. Όταν συντάξαμε τις τροπολογίες αυτές δεν ξέραμε ποια θα είναι η τελική απόλυξη, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Για τον πρώτο συμβιβασμό είναι ένα συμβιβασμός που επιτρέπει που επιτρέπει να συνδυάσουμε τη στρατηγική 2020 με τους βασικούς τρεις στόχους που εναπόκεινται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας εκπαίδευση, υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσης για τους νέους μας, απασχόληση και καταπολέμηση της στόχιας. Ο δεύτερος συμβιβασμός είναι ένα συμβιβασμό που βρήκαμε με τον Ξάμπα και που μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι έγινε στον προηγούμενο προγραμματισμό, διότι στον προηγούμενο προγραμματισμό, από, λόγω της κρίσης, χρειάστηκε να εισάγουμε ένα μέσο εμπελιξίας που επιτρέπει τον επαναπρογραμματισμό. Αυτό το λέγαμε στον συμβιβασμό Β και ευχαριστώ τον Τσάμπα όρι που δέχθηκε αυτόν τον συμβιβασμό. Συμβιβαστική γάμα σε υπάρχει μία διόρθωση. Όταν επιμένουμε εμείς αυτό το φάκελο του 25% που θα πρέπει να διατηρηθεί για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αυτό δεν θα πρέπει να υπολογιστεί μόνο βάση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά συνολικά όλου του φακέλου της πολιτικής συνοχής, έτσι όπως προτάθηκε από την Κομισιόν. Και η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν είναι μόνο το θέμα της κοινωνικής ε, το θέμα της κοινωνικής, ε, των κοινωνικών επενδύσεων αλλά και της πρακτικότητας. Μετά έχουμε έναν άλλο συμβιβασμό πολύ σημαντικό διότι εδώ διορθώνουμε την γλώσσα μας. Μιλάμε εμείς για το Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης το οποίο απειλείται ιδιαίτερα από το Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων κρατών που χρησιμοποίησαν παραδειγματικά στο παρελθόν του τα κονδύλια αυτού του ταμείου ή που τα χρησιμοποιούν ακόμη σήμερα από αυτό το πνεύμα. Αναγνώριση λοιπόν επί της ουσίας δηλαδή για την επάνωδο στην απασχόληση ε, των εργαζομένων που πλήττονται από την αλλαγή των αγορών εργασίαν και επίσης αναφερόμαστε εδώ στον τύπο των θέσεων απασχόλησης που, μιλάμε, που αναφέρουμε εδώ στη μεταβατική περίπτωση. Πολλές φορές γίνεται εξέταση αναπερίπτωση, αλλά οι καταρτήσεις οι οποίες είχαν προταθεί δεν ήταν απαραίτητα το καλύτερο, ε, το καλύτερα συμβατό με την εξέλιξη της αγοράς εργασίας. Αυτού του είδους η κατάρτιση θα πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους μας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, αηφόρο ανάπτυξη κλπ. Έχουμε την πέμπτη τώρα τροπολογία που αφορά στο μέλλον του προγράμματος βοήθεια προς τους ε, φτωχότερους. Όπως ξέρετε μετά από την απόφαση του δικαστηρίου παίζεται η επιβίωση αυτού του προγράμματος. Τα σχόλια τα οποία έχουμε από την Κομισιόν μας οδηγούν να σκεφτούμε ότι η επισητιστική βοήθεια θα, είναι, θα, θα, ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα. Δεν θελήσαμε εμείς να αποθαρρύνουμε την Κομισιόν τον προσανατολισμό, αλλά θυμήσαμε ότι η επισητιστική βοήθεια θα πρέπει να εντάξεται στο πρόγραμμα. Τροπολογία 6 Πρόκειται για μία τροπολογία που είναι χρήσιμη. Μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε τη δουλειά μας ως βουλευτές. Στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών, οι φιλελεύθεροι ζήτησαν να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και από αυτό το πνεύμα εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι βουλευτές να παρακολουθούν τη χρήση των κονδυλίων μέσα από τις επιτροπές παρακολούθησης. Η τροπολογία 7 πρόκειται για μια τροπολογία που αφορά στην νομοθετική πλευρά του κειμένου για τη διαθεσμική συμφωνία που θα συνοδέψει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελεί τη συνέχεια της ε, ε, γραμμής που συζητήσαμε με τη Μαριάν Άρκιν σχετικά με το μέλλον του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και εδώ αναφερόμαστε όμως πιο συγκεκριμένα στα μέτρα για τους γεωργούς και οι τροπολογίες μας επιτρέπουν να κάνουμε συμβιβασμούς γύρω από αυτά τα σημεία. Ο τελευταίος συμβιβασμός συμπεριλαμβάνει μια πολύ χρήσιμη πρόταση του Τσάμπα Όρη σχετικά με τον τρόπο χρήσης και τις προθεσμίες χρήσης αυτού του ταμείου και για το πώς εμείς επανεπενδύουμε το χρήμα το οποίο δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Και αυτό βάσει των αρχικών ποσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι εμείς έπρεπε να παρέμβουμε επί των ποσών γιατί φοβηθήκαμε εξάλλου ότι αυτό θα θεωρόταν απαράδεκτο. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά όταν έχουμε αυτές τις ανταλλαγές απόψεις στην Επιτροπή μας, να μπορούμε να προσεγγίζουμε όλες τις ε, ουσιαστικές πλευρές του, του, ζητήματος και να μην λέμε απλώς ότι οι ισχυώδεις εισηγητές τα βρήκαν μεταξύ τους. Ο Τσάμπα όρι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. διευκολύνατε την εργασία των σχεδόν εισηγητών με την καταπληκτική εισαγωγή σας. Από πλευρά ε, του ΕΛΚ ε, ε, δηλώνουμε ικανοποιημένοι, διότι ως επιτοπλίστων συμπεριλήφθησαν οι τροπολογίες μας στο τελικό σχέδιο. Μία ερώτηση έχω μόνο για την τροπολογία H. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένα ποσά, αλλά αν Τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει 429 εκατομμύρια για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Για ποιο λόγο εμείς θα πρέπει να το δεχθούμε. Πρόκειται για αποθεματικό και όλοι το γνωρίζουμε. Επίσης, άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι ε, εκείνο της ε, διεύρυνσης ε, του πεδίου εφαρμογής ε, και των πιο συγκεκριμένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας αυτού του ταμείου. Μα έχουμε μειώσει το κονδύλι. 500 εκατομμύρια ήταν αρχικά, αν θυμάμαι καλά. Εγώ θα πρότεινα να εισηγηθούμε διατήρηση του κονδυλίου. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, για μείωση. Και εξάλλου θα πρέπει να φροντίσουμε και τη διαπραγματευτική μας θέση για το μέλλον, διότι είναι θέμα που θα μας απασχολεί σε αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Άρα εμένουμε στο ποσό των 500 εκατομμυρίων. Αφήστε που είναι και θέμα αρχής παρότι δεν απορροφήθηκαν και τα 500 εκατομμύρια σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι στιγμής. Επίσης, θα θέλαμε να υποστηρίξουμε ε, γενικότερα τη γνωμοδότηση. Ακούγονται καλά τα ελληνικά, παρακαλώ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. No. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο να απαντήσω στον Τσάμπαρη. Ε, εγώ λέω ότι η λύση δεν είναι να βάλουμε νούμερα. Πρέπει να βάλουμε μία παρένθεση με τρεις τελίτσες. Διότι η θέση της Κομισιόν θα είναι να απορρίψει και τους Γιωργούς και το θέμα της ε, και την, ε, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ο στόχος μας δεν είναι 500 εκατομμύρια. Εμεί θέλουμε να πάρουμε πίσω όλο το χρήμα για να καλύψουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους γεωργούς κτλ. Πρόκειται για μια διαπραγμάτευση που πρέπει να μας πάει πέρα από τα 500 εκατομμύρια. Αν εμείς πούμε απλώς θέλουμε 500 εκατομμύρια, μα αυτό αντιφάσκει με τη θέση που εμείς θα λάβουμε για τους γεωργούς. Και αυτό, αυτή είναι η ανησυχία μου. Διότι 500 εκατομμύρια είναι αν εμείς μείνουμε περιοριστούμε στην πρόταση της Κομισιόν. Εμείς θέλουμε όμως να αλλάξουμε το φύλλο πορείας της Κομισιόν. Και ξέρω ότι αυτό κάνει και η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση δεν βάζει νούμερα. Βάζει χ. Μεγάλα χ, μικρά χ, τελίτσες, ό,τι θέλετε. Αλλά εγώ προτείνω να δεχτείτε αυτή την πρόταση. Τι λέτε. μου φαίνεται πιο λογικό όντω, Πρόεδρε. εάν ε, προτιμάτε να μην μιλήσουμε για συγκεκριμένα ποσά, ας μην μιλήσουμε για συγκεκριμένα ποσά. Είναι ίσως μια καλύτερη ιδέα. Ε, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι θα δημιουργηθεί προηγούμενο αν δεν μιλήσουμε για συγκεκριμένα ποσά. Ας βάλουμε αποσιοποιητικά ή ας βάλουμε παρένθεση και το βλέπουμε τελικά αυτό το ζήτημα, αυτό θα πρότεινα. Τέλεια λέει η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ και θα ψηφίσουμε. Τι γνωμοδότησή μας αύριο θα έχουμε μία μακρά συνεδρίαση ψηφοφορίας και η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα ψηφίσει 10 και 11 Οκτωβρίου. Σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Το λόγο έχει η κυρία Κορνέλισεν για την εξέταση των τροπολογιών στην έκθεσή της για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2012, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. 90 τροπολογίες είχαμε περίπου για τη γνωμοδότησή μου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους τις υπέβαλαν για τη συμβολή τους ως επιτοπλίστων ήταν ε, χρήσιμες ε, και θα βελτιώσουν ε, σε μεγάλο βαθμό την γνωμοδότηση. Και ξέρετε, οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ υπέβαλα το μεγαλύτερο αριθμό τροπολογιών, διότι ήμασταν περιορισμένες από τον αριθμό των λέξεων που μπορεί να ενέχει μία γνωμοδότηση και θέλουμε να τα πούμε όλα, θέλουμε να πούμε τόσο πολλά περισσότερα Άρα ε, το έκανα μέσω τροπολογιών. Ε, έγινε μια σύσκεψη για τις συμβαστικές τροπολογίες και εγώ κρίνω ότι ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και χρήσιμη η σύσκεψη αυτή, διότι οι περισσότεροι συμφώνησαν για τα περισσότερα. Συμφώνησαν σχεδόν για τα πάντα όλες οι πολιτικές ομάδες. Ένα κανθόδες ε, σημείο ήταν η παράγραφος που φέρει από των μισθών. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αποσιοποιήσουμε ε, ε, αυτό το θέμα και κρύβονται εδώ οι διαφορές ιδεολογικού περιεχομένου, διαφορές επί των αρχών ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες μεταξύ των οποίων και οι εξή. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει ή όχι το δικαίωμα να πει οτιδήποτε για τους μισθούς, ένα άλλο θέμα είναι αν ε, εκείνοι ισχυριστούν από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουν δικαίωμα, πώ εμεί θα αντιδράσουμε. Ε, επίσης μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και ενδοκομματικές ε, έρηδες πέρα από τις διακομματικές διαφορές και είναι αδύνατο να το αποσιοποιήσουμε όπως σας έλεγα. Πάντως σίγουρα θα μας απασχολήσει στις μελλοντικέ μας συζητήσεις το ζήτημα και ευελπιστώ ότι τελικά θα καταλήξουμε στην, σε κάποια ευρέως αποδεκτή συμβαστική τροπολογία. Εξυπακούεται ότι θα έχουμε διαπραγματεύσεις και με την Επιτροπή Έκων σε σχέση με το τι θα συμπεριληφθεί μέσα στην τροπολογία αυτή. Κατόπιν ε, υπάρχει μία σειρά τροπολογιών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις συμβαστικές. Εγώ θα βάλω ένα ε, ε, θετικό πρόσημο μόνο στο κατάλογο ψηφοφοριών. Υπάρχουν και κάποιες που δεν με βρίσκουν σύμφωνες, κυρίως από τους συντηρητικούς και από την ΚΟΕ, διότι τείνουν να πηχούν μία πραγματικότητα που λίγαν αποκλίνει από τη δική μου πραγματικότητα, αλλά δεν πειράζει γιατί ούτε εκείνοι υπερψηφίζουν τις δικές μας τροπολογίες. Κυρία Πρόεδρε, ε, περιμένω με ανυπομονησία τις δικές σας παρατηρήσεις για την εκθεσή μου. Σας ευχαριστώ κύριος Μπακ. Oui, merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κορνέλισεν για τη δουλειά της και για τη συνεργασία. Όπως επίσης και, όπως επίσης και όλους τους άλλους συναδέλφους. Εγώ θέλω να αποσύρω αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Κορνέλησεν στην ε, τοποθέτησή σας. Εμείς ε, συναντηθήκαμε οι σήμερα το απόγευμα και όπως είπε και η κυρία Κορνέλησεν καταφέραμε να λύσουμε τα περισσότερα προβλήματα των συμβιβαστικών τροπολογιών. Μένουν ακόμη μερικά σημεία που πρέπει να ρυθμίσουμε για τον συμβιβασμό ε σχετικά με τους μισθούς. Συμφωνώ ότι υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Έχω λοιπόν την γνώμη ότι θα συμφωνήσουμε γύρω από αυτό το θέμα. Επίσης, εγώ σκέφτομαι ότι αύριο θα καταφέρουμε να συνεννοηθούμε για ένα κείμενο το οποίο θα τονίζει τη σημασία των εργαζομένων και των δικαιωμάτων. Ε, θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω Ε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ε, πρόκειται εδώ για τη συνέχεια των εργασιών που είχαμε στην αρχή της χρονιάς. Το σημαντικό θέμα, το σημαντικό μήνυμα το οποίο βγαίνει σήμερα από την Επιτροπή μας είναι ότι υπάρχει μία τάση σήμερα στην Κομισιόν η οποία ε, πραγματικά χειροτερεύει και πρόκειται εδώ για το θέμα των μισθών. Δεν θέλω να αναφέρω την α ή την β περίπτωση, αλλά όταν γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν με την Τρόικα προτείνουν στην Ελλάδα ο κόσμος να δουλεύει 11 ώρες ε, τη μέρα, 60 ώρες τη βδομάδα, δεν ξέρω αν αυτό πραγματικά διέπεται από το πνεύμα το οποίο είχαμε όταν εγκρίναμε εμείς ε, την εκθεσή σας. Και μετά έχουμε το θέμα της ε, διόρθωσης των μισθών, ε, της προσαρμογής των μισθών. Το κόστος της εργασίας και της προσαρμογής των μισθών δεν πρέπει να αποτελεί ένα κεντρικό ζήτημα ε, και εμεί αναφέραμε όλα αυτά στην αρχική έκθεση αλλά το θέμα της διάρθρωσης μεταξύ των προσανατολισμών που ορίζει η Κομισιόν και των όρων που ισχύουν για τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στα κράτη-μέλη είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Τελευταία παρατήρηση. Αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική. Για το τι περιμένει δηλαδή η Κομισιόν για του χρόνου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να πει και αυτό τη γνώμη του για αυτό το εξάμεινο και σε αυτή τη φάση της διαδικασίας είναι να δούμε πώς η Κομισιόν έλαβε υπόψη της αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ως ουσιαστικό, γιατί λάβαμε την ετήσια έκθεση, την αναπτυξιακή έκθεση στην αρχή της χρονιάς και να ανασύρουμε μερικές διδασκαλίες ε, για του χρόνου. Η Κομισιόν ε, θα μας παρουσιάσει τις θέσεις της ε, για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης για το 2013. Θα έχουμε λοιπόν και εδώ ένα ε, στοχευμένο μήνυμα για το τι περιμένουμε από την Κομισιόν. Η κυρία Γεσλοβιέτσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια να βγάλει το όνομά μου από τον συμβιβασμό G. Διότι εγώ θα ήθελα να υποστηρίξουμε τις καινοτόμες λύσεις για την προστασία της απασχόλησης. Και θα ήθελα εδώ να αλλάξετε τη γλώσσα. Δεν θα ήθελα να μιλάτε εδώ για καταπολέμηση της ανεργίας, διότι εμείς ε, εδώ, ε, αν το πούμε αυτό, σκέφτομαι, έχουμε κατά νου τους ε, ανέργους. Αλλά εμείς εδώ μιλάμε για τον αγώνα για την απασχόληση. Μιλάμε για τα μέσα εκείνα τα οποία θα προωθήσουν την απασχόληση. Εγώ στην τροπολογία μου πρότεινα να μιλήσουμε για, αυτήν την, για αυτόν τον αγώνα για, υπέρ της απασχόλησης για το συμφέρον των νέων. Και αυτό γιατί το λέω. Διότι οι, είναι οι νέοι τελικά και οι γυναίκες ε, ε, ε, κάτω από τα 50 που χάνουν τις θέσεις εργασίας και μην μιλάμε μόνο για νέους. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια. Όλοι είστε ευχαριστημένοι. Η κυρία Κορνέλησεν. Ευχαριστώ όλους ε, τους σκιώδεις συζητητές για την υποστήριξή τους. Συμφωνώ και εγώ ότι ε, ελπίζω τελικά να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική ε, πρόταση και να έχουμε μια καλή γνωμοδότηση ε, την οποία θα μπορώ να παρουσιάσω στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων προς διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι ουσία του θέματος είναι η αξιολόγηση. Αυτό περιμένουμε εξάλλου για την επόμενη χρονιά. Και αυτό ε, προφανώς ε, υποστηρίζει την δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως υπογράμμισε και η κυρία Λουμπέκα. Και λυπούμεθα για το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταρτήσει εθνικά προγράμματα θέσεων απασχόλησης ε, παρότι έχουν δεσμευτεί για κάτι τέτοιο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου παρότι δεν τηρούν ούτε καν τις δικές τους υποχρεώσεις και τη δική τους ιδέα ουσιαστικά. Οπότε δεν καταλαβαίνω ποια κινητήριος δύναμη χρειάζεται για να δημιουργηθούν ε, θέσεις εργασίας ε, στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το σημείο. Προσπάθησα στην τροπολογία G να συμπεριλάβω ολόκληρη την αράδα της κυρίας Γιασλογιέκα σχετικά με τις ρηξικέλευτες λύσεις, διότι αυτές χρειαζόμαστε κατά τη γνώμη μου. Πιστεύω ότι διμερός και εκτός συνεδριάσεως θα ήταν καλύτερο να συζητήσουμε ή να διαπιστώσουμε αν τελικά χρειάζεται και είναι εφικτή και ευρέως αποδεκτεί μια επιπρόσθετη συμβαστική τροπολογία. Ουδάλλως προσμένω με ανυπομονησία στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μάλιστα, υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν θα προβούμε στην ψηφοφορία αύριο. Να μην ξεχάσουν οι συνάδελφοι τις ε, κάρτες τους για να ψηφίσουμε αύριο. Σημείο 10. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μογά Σαχτιέ για να ε, εξετάσουμε 233 τροπολογίες ε, για το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους ε, προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες, ε, δηλαδή τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεχίζεται η εργασία μετά την τήρηση της προθεσμίας με, μεταγραφή στην Εθνική Νομοθεσία του νομοθετήματος που ενέκρινε και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο ορίζει το οποίο ορίζει ε, την Αναβολή τη μεταφορά, αν θέλει, της οδηγίας το 2004 ε, για να ισχύσει μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2013. Άρα παράταση ισχύως εννοούσε μάλλον η ομιλήτρια. Την ε, περασμένη εβδομάδα συνεχίσαμε τον άτυπο διάλογο με την ε, Κυπριακή Προεδρία οποίος έλαβε χώρα παρουσία όλων των σχεδόν εισηγητών, όλων των πολιτικών ομάδων, τις οποίες είχαμε καλέσει για την ανταλλαγή απόψεων, όπως ακριβώς έγινε από την πρώτη ε, συνεδρίαση της ομάδας εργασίας μας, ε, με στόχο να συλλέξουμε το μέγιστο αριθμό πληροφοριών σχετικά με τις επιθυμίες των πολιτικών ομάδων. Όλοι μας ε, συμφωνούμε ότι βασικός στόχος είναι το να είναι άμεσα εφαρμοστέ η οδηγία, βρίσκοντας μία ισορροπία ανάμεσα ε, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνωτικά πεδία, αλλά ε, επιτυγχάνοντας ε, επίσης την απαιτούμενη ισορροπία με τρόπο ώστε να είναι δυνατές ε, οι εφαρμογές που απαιτούνται σήμερα κυρίως ως προς τον ιατρικό εξοπλισμό για το καλό της ε, δημόσιας υγείας. Προσπαθούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία όλοι από κοινού. Το κείμενο του Συμβουλίου έχει μεταξελιχθεί σε σχέση με την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα το δικό μας έργο βασίστηκε επί την, της προτάσεως της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να το διευκρινίσω αυτό. Καλέσαμε τους εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων ε, για να καταλήξουμε όλοι μαζί από κοινού το Σεπτέμβρη ε, σε μια κοινή μεθοδολογία και να λάβουμε υπόψη το σύνολο των τροπολογιών που ε, υπέβαλαν οι πολιτικές ομάδες. Σας υπενθυμίζω ότι υπευλήθησαν τελικά 233 τροπολογίες, 52 από το ΕΛΚ, 29 από τους σοσιαλιστές, 15 από τους φιλελευθέρους, 91 από τους πρασίνους, 19 από τους συντηρητικούς και 9 από την ΚΟΑ. Ας οικοδομήσουμε λοιπόν από κοινού μία μέθοδο εργασίας που θα μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις τροπολογίες αφενός και αφετέρου να ομαδοποιήσουμε όλες οι συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη και τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται ε, στα νέα, στο νέο σχέδιο που ε, επεξεργάζεται τώρα το Συμβούλιο. Δύο άτυπες συζητήσεις ε, ανάμεσα Στου ε, στους ε, ε, εισηγητές και έναν εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου είχαν προβλεφθεί για τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών και θα ήθελα, Πρόεδρε, αν συμφωνείτε, να προγραμματίσετε δύο συζητήσεις στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προτού λάβει χώρα η ψηφοφορία με τρόπο ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ευθυγραμμιστούμε με όλους τους υπολείπους για τις τροπολογίες που τελικά θα ψηφίσουμε. Τον Οκτώβρη στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας ή αλλιώς τον Νοέμβρη μπορούμε να εξετάσουμε αυτές τις τροπολογίες με στόχο η τελική ψηφοφορία να λάβει η χώρα τέλη Νοεμβρίου. Ε, πιστεύω ότι με αυτές τις επιπρόσθετες συζητήσεις θα είχαμε το, τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε ακόμη και τριμερή διάλογο πριν τα Χριστούγεννα, αν συντρέξει λόγος. Ε, αυτά έχουν συμβεί μέχρι στιγμής. Προσπαθήσαμε να μην χάσουμε χρόνο και να κρατήσουμε την ίδια μέθοδο εργασίας ανταλλάσσοντας το μέγιστο αριθμό πληροφοριών και θέτω υπόψη των συναδέλφων ε, το σχέδιο, περιγράφοντας με αυτή την ε, σύνοψη ε, την μέθοδο εργασία μας, καθώς και την πρότασή μου για τις νέες συζητήσεις στην Επιτροπή Απασχόλης. Ευχαριστούμε, η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ την Μωρήν Σαρτιέ για την μέχρι τώρα δουλειά της. την εκτιμώ ιδιαίτερα μου είναι από τους πλέον συμπαθείς συναδέλφους. Χαίρομαι που εργάζομαι μαζί της. Αλλά ε, στεναχωριέμαι γιατί σήμερα πρέπει να μιλήσω λίγο διαφορετικά από ό,τι μιλάω συνήθως. Είμαστε σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο υπογραμμίζω. Δεν είμαστε στο Συμβούλιο, είμαστε στο Κοινοβούλιο το μοναδικό δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ ευαίσθητο και είμαστε εδώ σήμερα σαν να μην πέρασε ούτε μία ημέρα από όταν ξεκινήσαμε την εργασία μας για αυτό το θέμα, ενώ κοντεύει να περάσει ένας χρόνος. Και αυτό με στεναχωρεί με στεναχωρεί πάρα πολύ. Γιατί ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία, ε, πηγαίναμε χέρι-χέρι δουλεύοντας για, αυτό, για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση, φτάσαμε σε ένα σημείο και ξαφνικά σιγεία σειρμάτου. Τίποτα. Κουβέντα. Όντως κατετέθησαν οι τροπολογίες. Συνήθως όταν κατατίθενται τροπολογίες ποιο είναι το επόμενο βήμα δεν ξέρω μπορεί να κάνω λάθος περιμένουμε τις συμβιβαστικές δεν τις λάβαμε περνούσε ο καιρός περνούσε ο καιρός παράλληλα υπήρχε το θέμα ότι η οδηγία του 2004 κάποια στιγμή θα έλυγε πήγαμε στην παράταση του χρόνου εφαρμογής και ισχύως της οδηγίας του 2004. Πήγε 31 Οκτωβρίου του 2013. Κινδυνεύουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν δεν εργαστούμε γρήγορα, να μείνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι και οι Ευρωπαίοι ασθενείς χωρίς νομοθεσία. Και άρα πιεζόμαστε να τελειώνουμε με το θέμα αυτό σε πρώτη ανάγνωση. Για να τα σκεφτούμε όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Τι σημαίνουν για τον Ευρωπαίο πολίτη για λογαριασμό του οποίου εργαζόμαστε. Θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Μακάρι, γι' αυτό εργαζόμαστε όλοι εδώ. Για να βγει ένα καλό, ισορροπημένο αποτέλεσμα. Υπάρχει λοιπόν το Κοινοβούλιο. Υπάρχει και το Συμβούλιο. Το ξέρουμε και αυτό το Συμβούλιο το έχουμε δει επανειλημμένα να εργάζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αποσιοποιητικά. Δηλώνω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Κυπριακή Προεδρία. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ο χρόνος που έχει χαθεί και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε χειριστεί το θέμα με στεναχωρεί, δεν με ικανοποιεί άκουσα την κυρία Σαρτιέ η οποία ζητούσε άλλες δύο συζητήσεις όχι άλλες δύο, άλλες 102 συζητήσεις να κάνουμε αν πρόκειται να καταλήξουμε για το καλό του Ευρωπαίου πολίτη. Αλλά το θέμα, είναι, το θέμα έχει δύο διαστάσεις. Πρώτον, να συζητάμε επιπίου θέματος, όταν ήδη δεν έχουμε τίποτα μπροστά μας, στη διάθεσή μας. Όταν περιμέναμε έναν εμπειρογνώμονα να έρθει εκ μέρους του Συμβουλίου και να μας πει πού ακριβώς άλλαξε και πού βαδίζει το Συμβούλιο και χάθηκε στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ο ειδικό. Δεν τον είδαμε ποτέ. Εξαϊλώθηκε, εξαερώθηκε, εξαφανίστηκε. Να πάμε λοιπόν σε άλλες δύο συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, σε 102. Αλλά ταυτοχρόνως είναι και η προθεσμία. Τι θα γίνει, πού θα οδηγηθούμε. Εν πάση περιπτώσει τα περιγράφω όλα αυτά για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, για να μην ωραιοποιούμε καταστάσεις και για να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Μπροστά μας λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχουμε μία προθεσμία που μας πιάνει από το λαιμό. Μπροστά μας έχουμε την απόλυτη επιτακτική ανάγκη να ξαναδούμε τα όρια, τα, τα οποία πρέπει να υπάρχουν στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μπροστά μας έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι κάθε μέρα κινδυνεύουν είτε μέσα στα νοσοκομεία είτε αυτοί που εργάζονται στα ζητήματα του στρατού και μπροστά μας έχουμε ασθενείς που κινδυνεύουν να πεθάνουν εάν δεν μπουν να κάνουν μία μαγνητική τομογραφία. Όλα αυτά πρέπει να τα εξισορροπήσουμε και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ήδη εμείς ως σοσιαλιστές έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και είναι κρίμα να κάνουμε αυτού του είδους τη συζήτηση τώρα, όταν ήδη οι προτάσεις μας είναι πολύ κοντά με αυτές που είχε καταθέσει αρχικά η κυρία Σαρτιέ. Άρα δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκπτώσεις. Πρέπει να πάμε μπροστά τη δουλειά μας, έχοντας στο μυαλό μας να εξυπηρετήσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη και, συγγνώμη που το λέω συνάδελφοί μου καλή, όχι το Συμβούλιο. Δεν με ενδιαφέρει το Συμβούλιο. Με ενδιαφέρει ο Ευρωπαίος πολίτης. Δεν με ενδιαφέρουν οι τύποι. Με ενδιαφέρει η ουσία. Ε, είμαι εδώ. Είμαι στη διάθεση της εισηγήτριας για άπειρες συζητήσεις, νυχθημερών να εργαστούμε, αλλά να ξέρουμε πού πάμε. Να ξέρουμε επί ποιου εδάφους περπατούμε και εν πάση περιπτώσει το συμβούλιο να καταλάβει ότι υπάρχει ένα κοινοβούλιο επαναλαμβάνω το μοναδικό δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο της ευρωπαϊκής ένωσης και οφείλει να το λαμβάνει υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη από όλους και από όλες εάν υπήρχε μια ένταση στον τρόπο της εκφοράς του λόγου μου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ η κυρία Χάρκιν τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Σατία ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ισορροπία ανάμεσα στην έκθεση των εργαζομένων στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αλλά και τις απαιτήσει για κάποιες αποκλήσεις σχετικά ε, με διάφορες ιατρικές ε, εφαρμογές ε, όπως η τομογραφία. Ε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε συναντήσεις ε, με την κυρία Σαρτιέ, τους ε, Σκιώδης και το Συμβούλιο με ακούσαμε για τι προόδου που έχουν σημειωθεί, συγκεκριμένα τεχνολογικέ και επιστημονικέ προόδου που έχουν σημειωθεί. Η διεθνή Επιτροπή για τις Μη του Ακτινοβολίες έχει κάνει κάποιες εισηγήσεις, οποίε οφείλουμε να λάβουμε επίση υπόψη. Ε, συμφωνώ και με την κυρία Ράπτη, είναι ε, καθοριστική σημασία ο παράγοντα χρόνο, ε, και αν κατάλαβα καλά είπε ότι δεν την νοιάζει τι κάνει το Συμβούλιο. Μα όμω θα τη έλεγα ότι θα πρέπει παρόλα αυτά να καταλήξουμε στη συμφωνία με το Συμβούλιο και άρα θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια ισορροπία εν τέλει. Νομίζω ότι αυτό που μας προτείνει η συγγήτρια είναι ένα συμβασμός που θα μπορούσε τελικά να λειτουργήσει και συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστό το Κοινοβούλιο, αλλά αυτό είναι το, η δική μας δουλειά. Στους τριμερείς διαλόγους σας ερημνήσουμε τόσο ώστε να έχει το σεβασμό που το αξίζει το Κοινοβούλιο. Ε, θα πρέπει να βρεθεί μια συμφωνία ανάμεσα στι ε, προτάσεις ε, που υπάρχουν επιτάπητο ε, και τις δικές μας τροπολογίες. Ε, νομίζω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή είναι η καλύτερη ρότα που έχουμε να ακολουθήσουμε. Μιλήσατε για τις ε, συζητήσεις στην Επιτροπή. Βεβαίως, συμφωνώ. Τώρα αν θα είναι δύο ή περισσότερες θα το δούμε. Πιστεύω ότι οι ισχυώδεις εισηγητέ πρέπει να εργαστούν σε επιτοπλίστων για την επεξεργασία των συμβαστικών τροπολογιών. Αυτή είναι η κατάσταση προς το παρόν και αυτό είναι το χρονικό χρονοδιάγραμμα που έχουμε και δοθέντων όλων αυτών θα συμφωνήσω με τις προτάσεις της για την ε, περαιτέρω πορεία μας, ε, Πρόεδρος. Θέλει κανεί άλλο το λόγο, πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Μα, μόλις μιλήσατε, κύριε Ράπτη. Κρινήσω μόνο, κυρία Πρόεδρε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, δεν εννοούσα ότι δεν με νοιάζει ποια είναι η γνώμη του Συμβουλίου τι λέει το Συμβούλιο, τι προτείνει το Συμβούλιο. Ασφαλώς και με νοιάζει, ασφαλώς και έχω στο μυαλό μου πρώτα και κύρια την επίτευξη συμφωνίας. Αυτό είναι η επιδίωξη της εργασίας μας. Όταν λέω ότι δεν με νοιάζει τι κάνει το Συμβούλιο, εννοώ από πλευράς χρόνου τον οποίο διαχειρίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Προφανώς και δική μου επιδίωξη όπως και όλων μα είναι να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατό συμβιβασμό. Ενδεχομένως δεν εκφράστηκα εγώ σωστά. Ζητώ συγγνώμη αν δεν έγινα κατανοητή. Ευχαριστώ. Merci. Donc, il δεν θέλει το λόγο. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν και μετά στην εισηγήτρια, να πω και εγώ μερικά πράγματα. Θα πρέπει η εισηγήτρια να μας διευκρινίσει αυτές τις δύο περαιτέρω ανταλλαγές απόψεων στην Επίτροπη, γιατί εμένα ξέρετε δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι λένε σε κάθε, η αυταρέσκεια σε κάθε Επίτροπη, όπου οι και εισηγητές από το συγχαίρονται για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων. Εδώ στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στις ακτινοβολίες και τέρμα. Συγγνώμη που είμαι απότομη. Από πίσω υπάρχει ένα τεράστιο λόμπι και ιατρικό αλλά και κατασκευαστών αυτού του υλικού που δεν θέλουν καν να ακούσουν να μιλάμε για αυτή την νομοθεσία. Γι' αυτό έχουν μπλοκαριστεί τα πάντα στο Συμβούλιο. Γι' αυτό υπήρξε και η αναβολή της έγκρισης της προηγούμενης οδηγίας και γι' αυτό η θέση που θα εγκρίνουμε εμείς είναι σημαντική. Τώρα, Είχε γίνει και η διαβούλευση με τους εργαζόμενους, μπορώ να φανταστώ γιατί δεν θυμάμαι ε, υπό ποιους όρους έγινε. Αλλά όταν ακούω εγώ τους εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου, εντάξει, αλλά να ακούσουμε όμως τι λένε και εμπειρογνώμονες του Διεθνούς, του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας. Ε, να ακούσουμε και άλλους ε, για να ισορροπήσουμε τις θέσεις. Και τώρα να θέσω και μία αθώα ερώτηση. Αφελή. Εμείς έχουμε 211 τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι. Δηλαδή, πριν σταματήσουμε την διαδικασία, για να περάσει η παράταση της ε, υγείας. Τώρα, αντί να συζητάμε και να ξανασυζητάμε στην Επιτροπή, εδώ αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να ξανανοίξουμε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και να μπορέσουμε να βρούμε και το σωστό συμβιβασμό στα παρασκήνια. Δεν είμαι σίγουρη, εγώ ερωτήσεις κάνω, έτσι μου περνάνε από το κεφάλι. Και ε, αν περνάνε βέβαια όλα αυτά από το κεφάλι μου, μπορεί να περνάνε και από το κεφάλι αλλωνών. Έχουμε εδώ 233 τροπολογίες, σαν να μην έχει μεσολαβήσει τίποτα από το Δεκέμβριο του 2011. Και στο τέλος, αυτό το οποίο φοβούμε είναι ότι το μόνο το οποίο θα έχουμε μπροστά μας ως επιλογή είναι να εγκρίνουμε την κοινή θέση που θα περάσει από το Συμβούλιο. Εγώ εδώ θέτω ένα μεθοδολογικό ζήτημα λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή την ε, διαδικασία σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και τη δυσκολία της συζήτησης στο Συμβούλιο. Για να απαντήσουμε όμως όλα αυτά τα ερωτηματικά, θα μας διαφωτίσει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και μετά η εισηγήτρια θα μας πει και αυτή πώς θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι η κατάσταση είναι αρκετά πολύπλοκη, δηλαδή το Συμβούλιο ξεκίνησε την ανάλυση εκ παραλίλου και ξα... ξανάφτιαξε το κείμενο από την αρχή, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2011 και μετά. Στο Συμβούλιο τα πράγματα εξελίσσονται καλώς και χωρίς εγώ να θέλω να υποκαταστήσω τους του Συμβουλίου, Πιστεύω ότι το Συμβούλιο θέλει να εγκρίνει ένα general approach, μια γενική συμφωνία για τις αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό θα γίνει αν στην ομάδα αύριο για τις κοινωνικές υποθέσεις μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τα δύο-τρία μικροσημεία τα οποία εκκρεμούν. Στις 4 Οκτωβρίου, αν συμβούν όλα αυτά, θα έχετε ένα κείμενο το οποίο θα σας διαφωτίζει για την ε, διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε, άνοιγμα προθεσμίας τροπολογιών κλπ. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μία λύση. Και αυτό λόγω του λίγου χρόνου που έχουμε μπροστά μας. Θέλω όμως να σας διασφαλίσω ότι να σας διασφαλίσω για αυτά τα οποία αποφάσισε η Κομισιόν τον Ιούνιο του 2011. Εμείς αλλάξαμε πορεία σε μεγάλο βαθμό και αλλάξαμε πολλά πράγματα, αλλά μετά επανήλθαμε στο αρχικό κείμενο της Κομισιόν. Δεν ήταν ιδιαίτερα εύπεπτο βέβαια αυτό το κείμενο. Αλλά οι αρχές που βρίσκονται στη βάση της πρότασης υπίστανται και στο κείμενο το οποίο κυκλοφορεί στο Συμβούλιο. Και αυτό είναι ένα καλό νέο. Βέβαια μερικά πράγματα δεν είναι πια τόσο ριζοσπαστικά όσο στην πρώτη πρόταση της Κομισιόν, αλλά... Αλλά Η Κομισιόν πρόσεξε ιδιαίτερα το πρόβλημα του ιατρικού κλάδου και της δυνατότητας που πρέπει να έχει ούτως ώστε να θεραπεύει τους ασθενείς. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στην τωρινή πρόταση. Το ίδιο ισχύει και αυτό το οποίο προτείναμε για το στρατό, τότε για το ΝΑΤΟ ήτανε, όταν μιλούσαμε για, στρατηγική, για δραστηριότητες. Και είχαμε και ένα παράθυρο για συγκεκριμένες περιπτώσεις, για να επιτρέψουμε δηλαδή μερικές παρεκκλήσεις για τη βιομηχανία. Αυτά θα συζητηθούν αύριο. Εμείς πρέπει να προσέξουμε ε, την προστασία των εργαζομένων. Οι παρεκκλήσεις, οι εξαιρέσεις θα πρέπει να δίνονται μόνο σε ιδιάζουσες περιπτώσεις, όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο άλλαξε ουσιαστικά. Είναι πολλά σημεία για τα οποία διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να δώσουμε κατευθύνσεις ε, για την εφαρμογή υγείας και για το Συμβούλιο προσέθεσαν στο άρθρο 13 μερικά πράγματα ε, ε, στον οδηγό των καλών πρακτικών. Πρόκειται εδώ για τη τεχνική εφαρμογή ορισμένων πλευρών, ούτως ώστε ο καθένας να καταλάβει τι κρύβεται από πίσω. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν διαγραφεί από τα παραρτήματα, τα ξαναβρίσκουμε στο κόρπους του κειμένου. Ε, είναι ένα έγγραφο ιδιαίτερα συνεκτικό και οι τροπολογίες δεν αναφέρονται που έχετε εδώ, δεν αναφέρονται λοιπόν σε αυτό το κείμενο γιατί πολλά από τα μέλη της Επιτροπής σας θα βρούνε τη θέση τους μέσα σε αυτό το κείμενο. Αυτά κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, θέλω να πω ότι έξω από εδώ δεν είναι ιδέα μου εγώ να, να, να, παρατείνω τις ε, ε, προθεσμίες. Αλλά μιλάμε εδώ όμως για το άνοιγμα της διαδικασίας, επανάνοιγμα της διαδικασίας για την κατάθεση τροπολογιών. Διότι έχουμε εδώ μια εντελώς καινούργια διαδικασία. Εμείς έχουμε τη θέση μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο προχωρήσαμε και περιορίσαμε και κοντίναμε και την χρονική προθεσμία που είχαμε με το Συμβούλιο. Δεν είμαστε εμείς που θα τα καθυστερήσουμε. Λοιπόν, πολλά πράγματα, πολλές από αυτές τις τροπολογίες μπορεί να καλύπτονται από το νέο κείμενο, αλλά προσθέτω ότι εγώ θα δυσκολευτώ ιδιαίτερα να ψηφίσω αυτό το κείμενο, άμα δεν ξέρω σαφώς υπό ποιους όρους προστατεύει αποτελεσματικά τους εργαζόμενους του κλάδου, διότι αυτός είναι ο στόχος του κειμένου και όχι δηλαδή το να ξέρουμε αν οι κατασκευαστές αυτών των μηχανημάτων ή οι γιατροί είναι ευχαριστημένοι από τον συμβιβασμό του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προστασία των εργαζομένων που είναι αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής. Κυρία Μωγάν Σαντιέ, τώρα για να μας μιλήσει για τις δύο επόμενες συσκέψεις και για να κάνει τη σύνεψη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, άκουσα ε, τους ε, συναδέλφους. Ε, λυπάμαι που η κυρία Ράπτη δεν ήρθε στην τελευταία συνεδρίαση που έγινε για τους εισηγητές. Θα μπορούσε εκεί να τοποθετηθεί και σίγουρα θα πρέπει Αυτά που είπατε για το Κοινοβούλιο, ότι είμαστε δημοκρατικά εκλεγμένοι και είμαστε το πρώτο θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί του πολίτε, ε, δεν νομίζω ότι ισχυρίζεται κανεί το αντίθετο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποια πράγματα να μα παθιάζουν, αλλά ασχοληθούμε καλύτερα με τα πράγματα ε, που έχουν σημασία, δηλαδή με την ουσία τη έκθεση, διότι όλοι θέλουμε να προχωρήσει. Δεύτερο σημείο ούτε δεν θα έπρεπε ε, να, να μου προσάπτουν ότι παρατείνω εγώ τις ε, ε, προθεσμίες, διότι πιστεύω ότι ενεπλάκην ικανοποιητικά στις συζητήσεις με το Συμβούλιο και ελήφθη αυτή η απόφαση παράταση όχι κατά δύο χρόνια αλλά 18 μήνες, διότι ήταν απαραίτητο και προσπαθούμε συντεταγμένα να προχωρούμε και έτσι λαμβάνουμε και τις αποφάσεις μας ε, οπότε προτείνω ε, ε, αθρώα προσέλευση στις εσκήψεις για να μην έχουμε άγονες συζητήσεις στην Επιτροπή. Πρόεδρε, εγώ αυτό επιθυμώ. Το πρόβλημα που καλούμεθα να επιλύσουμε έχει δύο όψεις. Ε, πρώτον, όντω ε, εξυπακούεται ότι εργαζόμαστε για να προστατεύσουμε την υγεία των εργαζομένων. Αλλά κάποια στιγμή ε, όλοι χρειάζονται ιατρικές εξετάσεις. Δεν το εύχομαι σε κανέναν να χρειαστεί ε, τομογραφία για οποιοδήποτε όγκο γνωρίζετε ε, κυρία Ράπτη ότι δεν το εύχομαι σε κανέναν αλλά όταν χρειάζεται θα πρέπει κάποιο να έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί ε, αλλά α μην λειτουργούμε δημαγωγικά και να ξέρουμε ότι ανάμεσα στην υγεία των ασθενών και την υγεία του συνόλου των συμπολιτών μας θα πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή, μια μέση λύση και α μην αρχίσουμε να μιλάμε για τα προβλήματα που προέρχονται από τη βιομηχανία βιομηχανία, διότι είναι το θέμα τη Ευρωπαϊκή ηθαγένεια ουσιαστικά και των δικαιωμάτων που συνεπάγεται. Εγώ έτσι προσεγγίζω το θέμα και ε, μέσα αυτή τη λογική θέλω να κινούμε. Η δεύτερη όψη του προβλήματος ε, με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι έγκυται στο εξή. Ε, με το πέρασμα των διαδοχικών προεδριών, οφείλω να το ομολογήσω και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει αλλάξει σημαντικά το κείμενο ε, σε σχέση με την αρχική πρόταση. Σήμερα λοιπόν πρέπει αυτό το χάσμα ανάμεσα στο αρχικό κείμενο και το τελικό να το καλύψουμε με τον πλέον επικοδομητικό και παραγωγικό τρόπο. Όντως, ε, δύο είναι οι τρόποι για να το πετύχουμε αυτό, είτε και να πω παρενθετικά ότι δεν είμαι υπέρ των ατερμών συζητήσεων και των αγώνων συζητήσεων. Είτε λοιπόν θα αρχίσει να τρέχει η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, γνωρίζοντας ότι θα ε, κινηθούμε μέσα σε ένα εξαιρετικά αυστηρό χρονοδιάγραμμα, είτε θα συνεχίσουμε ε, τις συζητήσεις μας για τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εάν ανοίξουμε και πάλι, ε, κινήσουμε και πάλι την διαδικασία υποβολής τροπολογιών, τι θα γίνει με τις ήδη υποβληθήσεις τροπολογίες. Αυτή είναι η μοναδική ερώτηση που έχω δεν έχω καμία ένσταση. Ε, ας ε, επανεκκινήσει η διαδικασία, αλλά ε, προσοχή στο χρόνο διότι, και προσοχή στις προηγούμενες τροπολογίες, διότι εν τέλει αν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο που απηχεί την άποψη σύσσωμου του Κοινοβουλίου και ε, η Ρίστο εν παρόδο, η κυρία Ράπτη, είναι μέσα στα μελήματά μου να είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Θα πρέπει λοιπόν να ε, σεβαστούμε τον ε, απότερο στόχο σε σχέση με τις εργασίες όλων των θεσμικών οργάνων και σε σχέση με τους δικούς μου στόχους. Οπότε ξαναρωτάω, Πρόεδρε, τι θα γίνει με τις ήδη υποβληθείς τροπολογίες αν επανεκκινήσει η διαδικασία. Η κυρία Ράπτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν σωστά αντιλαμβάνομαι, έχουμε μπροστά μας ένα νέο κείμενο βάσης, διότι από αυτά που άκουσα και από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, αλλά ακούγοντας και την κυρία Σαρτιέ να μιλάει για ένα χάσμα ανάμεσα στο παλαιό κείμενο και το καινούριο, αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να εργαστούμε εκ νέου πάνω σε τροπολογίες, πάνω σε ένα καινούριο κείμενο. Ε, υπό αυτήν την έννοια, η πρότασή σας να ξαναξεκινήσουμε τη διαδικασία ε, μου μοιάζει λογική. Φαίνεται απολύτως λογική. Παράλληλα, θέλω να σημειώσω και να υπενθυμίσω ότι στην εργασία που έχουμε κάνει με την κυρία Σαρτιέ ε, έχουμε φτάσει, είχαμε φτάσει, είχαμε φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο α, να, ε, συναντιόντουσαν οι απόψεις μας σε ένα πολύ μεγάλο όγκο της εργασίας μας. Αλλά από τη στιγμή που το κείμενο βάσης του Συμβουλίου έχει αλλάξει, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε όλο το έργο αυτό ε, λαμβάνοντας υπόψη και τα χρονικά περιθώρια, λαμβάνοντας υπόψη και την αναγκαιότητα, όπως και εγώ είπα και νομίζω στο, καθενό καθενός στο μυαλό υπάρχει, ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα, αλλά να λυθεί σωστά, ε, βλέπω ε, να είναι μια λογική λύση η επανεκκίνηση της διαδικασίας Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτά τα θέματα χρονοδιαγράμματος Συνήθω, δηλαδή α το πω αλλιώ, δεν ήθιστε στην Επιτροπή να τα ρυθμίζουμε αυτά και λυπάμαι που δεν ήμουν ενημερωμένη ήδη για να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να μην κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσει εδώ στην Επιτροπή. ούτω ή άλλω δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες συζητήσει. Τέλος πάντων, ε, ε κυρία Σαχή, ε, δεν ε, μου, μου δώσατε την εντύπωση ότι απαντήσατε για αυτό που σας ρώτησα. Τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε σε αυτές τις δύο επιπρόσθετες συσκέψεις που ζητάτε να διοργανωθούν. Ε, θα προτιμούσα να με είχατε ενημερώσει ε, πρώτη συσκέψη της Επιτροπής μας για να ε, είχαμε αποφύγει όλη αυτή την συζήτηση. Απάντηση, Πρόεδρε. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στη συζητήση με το Συμβούλιο με, μια, με ένα, ε, πώς να σας το πω, ε, κρατεό αποτέλεσμα ψηφοφορίας, μια ισχυρή πλειοψηφία για να περάσουμε ένα θετικό μήνυμα στο Συμβούλιο. Αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε συμφωνήσει επί ενός συγκεκριμένου αριθμού συμβαστικών τροπολογιών, ούτως ώστε να είμαστε συσπηρωμένοι. Αυτές ε, οι συμβαστικές ε, τροπολογίες αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, πρέπει όμως ταυτόχρονα όλα τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης να είναι ενήμερα για την πορεία των διαπραγματεύσεων αυτών με τους σκιώδεις εισηγητές. Και αυτό είναι το αντικείμενο των δύο συσκέψεων που σας προτείνω. Εάν των δύο συζητήσεων μάλλον. Εάν τώρα θέλετε να επανεκκινήσουμε τη διαδικασία και να υποβάλουμε όλοι οι τροπολογίες, αυτό θα αποφασιστεί από το σύνολο των μελών της Επιτροπής. Εμένα αυτό ε, που με ενδιαφέρει είναι να έχουμε ξαναλέω την ισχυρότερη δυνατή ε, πλειοψηφία ε, στην ε, ψηφοφορία που θα γίνει στην Επιτροπή Απασχόλησης, διότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με τους αμφιταλαντευόμενους. Δηλαδή σε μία διαπραγμάτευση πρέπει να ισχύσει μία σχέση εμπιστοσύνης, αλλά όχι μόνο να είναι και δεσμευτική η τοποθέτησή μας ε, σε σχέση με αυτά που θα πράξουμε στο μέλλον και εννοώ την ψηφοφορία. Πρόεδρος, επιθυμείτε να έχουμε δύο ανταλλαγές απόψεων πριν την ψηφοφορία. Μία για να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και την άλλη για ποιο λόγο απάντηση για την περίπτωση όπου θα σημειώνονταν αλλαγές μετά από την πρώτη για να είμαστε όλοι σύμφωνοι. Και συμπληρώνω, αν έχουν δεσμευτεί όλοι επαρκώς ε, και είμαστε σίγουροι ότι έχουμε μια ισχυρή διαπραγματευτική βάση, θα μας έφτανε και μία ανταλλαγή απόψεων, μία συζήτηση. Ε, το, ο απότερος στόχος μας είναι να μην αλλάξουμε τη θέση μας. Πρόεδρος, εγώ διαπιστώνω ότι μισή ώρα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα ενώ στην ημερήσια έχει προβληθεί προβλεφθεί εξέταση των τροπολογιών. Ε, εγώ τίποτα δεν έμαθα για την ουσία του φακέλου πάντως από αυτή τη συζήτηση και πραγματικά Ειλικρινά, ως πρόεδρος Επιτροπή Επιτροπής έχω μπουχτίσει με αυτέ τι συνεδριάσεις επιτροπών που τίποτα δεν μαθαίνω για ε, το περιεχόμενο των εκθέσεων και κρίμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και αύριο που θα έρθουν οι δημοσιογράφοι, ο τύπος, οι πολίτε οποιοδήποτε να με ρωτήσει «Μα τι λέγατε χθε, τι συζητούσατε» ε, λοιπόν δεν δίναμε ε, βγαίνοντα από αυτή τη συνεδρίαση να σα πω προ τα πού κατευθυνόμαστε και τι κάνουμε με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ. Θα μπορούσαμε δεδομένων των νέων στοιχείων ε, από το Δεκέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα δηλαδή. Και χωρίς να περιπλέξουμε ε, περίτα το έργο της ε, εισηγήτριάς μας, ας ορίσουμε μια πολύ σύντομη προθεσμία ε, υποβολής τροπολογιών για να συμπληρώσουμε το, πακέτο, το διαπραγματευτικό πακέτο μας. Δηλαδή, οι 233 τροπολογίες που είναι επιτάπητος παραμένουν ως έχουν. Οι των σκιωδών που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη διαπραγματευτική μας βάση δύναται να το πράξουν είτε στα αγγλικά είτε στα γαλλικά μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Αυτό μας επιτρέπει να διατηρήσουμε το ίδιο χρονοδιάγραμμα για τη συνέχεια των εργασιών μας. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε από αυτό παρακαλώ. αυτό καταδεικνύει ότι είναι ενδελεχής η εξέταση του ζητήματος από πλευράς μας ε, και λόγω της παράτασης ισχύω της οδηγία και δεδομένων των νέων στοιχείων να προτείνουμε νέα προθεσμία. Δεύτερον, εάν η συγγήτρια θεωρεί ότι μέσα σε αυτή την προθεσμία προλαβαίνει να συντάξει συμβαστικές τροπολογίες μέχρι τις 8-9 Οκτωβρίου, αυτό θα πρέπει να μου το πείτε αγαπητή Ελισάβετ, Εάν λοιπόν συμφωνείτε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες, εκτός και αν πρόκειται για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για ε, τις τροπολογίες, εν τη αυτή περιπτώση θα ε, διοργανώσουμε δεύτερη ανταλλαγή απόψεων σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο στις 19 Οκτωβρίου, ε, με μια ψηφοφορία που θα γίνει στις 28-29 Νοεμβρίου. Σας ικανοποιεί το χρονοδιάγραμμα, ε, κύριε Σαφτή. Επί της ουσίας, κυρία Πρόεδρε, εγώ μπορώ πάρα πολύ εύκολα να εξηγήσω στον καθένα από εδώ, που είναι εδώ παρόν, το περιεχόμενο των τροπολογιών. Τα προβλήματα που ανέφεραν οι διάφορες πολιτικές ομάδες, Είχαν μερικές μικροδιαφορές, αλλά όλοι είχαν το ίδιο βασικό πρόβλημα, το θέμα των παρεκκλήσεων. Σε ποιο βαθμό εμείς μπορούμε να έχουμε παρέκκληση σε μια, ε, επί μιας γενικής νομοθεσίας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Ιατρική παρέκκληση, αμυντική παρέκκληση. Αυτό είναι το πρόβλημα των παρεκκλήσεων. Δεύτερο σημείο για το οποίο υπάρχουν, υπάρχουν τροπολογίες είναι οτιδήποτε αφορά στις τιμές έκθεσης ή δράσης. Δηλαδή, πρόκειται για την ένταση των μαγνητικών, τις βαθμίδες μάλλον μαγνητικού πεδίου, στις οποίες μπορεί να εκτεθεί ένας εργαζόμενος. Μετά έχουμε τον κώδικα των καλών πρακτικών για να μπορέσουμε να πλησιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την προστασία της υγείας των, εργαζομένων, των εργαζομένων. Πολύ σύντομα. Ε, λυπούμε κυρία Πρόεδρε ε, που διαμορφώσατε την εντύπωση ότι δεν υπήρχε καμία πληροφορία επί της ουσίας. Μπορώ να σας τις αναλύσω όσο θέλετε. Και έχουμε και ένα σωρό τροπολογίες που έρχονται από διάφορες πολιτικές ομάδες και συγκλίνουν σε αυτά τα τρία προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα ουσίας τα οποία τίθενται και όλοι είμαστε πεπισμένοι, έχουμε το κίνητρο για να πετύχουμε αυτή την διαπραγμάτευση. Τώρα, για τις τροπολογίες, το χρονοδιάγραμμα με βολεύει απόλυτα. Αν δω ε, αν και οι συνάδελφοι, οι σκιώδεις έχουν την ίδια βούληση να καταλήξουν σε συμβιβασμό, Αυτό με βολεύει απόλυτα. Και να προχωρήσουμε με το τελικό χρονοδιάγραμμα που σας ανέφερα προηγουμένως. Είπα αυτού τους όρου. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ξανανοίγει μέχρι τι 25 Σεπτεμβρίου στι 12. Στα αγγλικά μόνο. Κυρία Πρόεδρε, εγώ ως εισηγήτρια ζητώ οι τροπολογίες να είναι αγγλικά και γαλλικά. Κυρία εισηγήτρια, αρχικά εγώ είχα σκεφτεί αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι αυτό δημιουργεί ανισότητα ως προς τα μέλη της Επιτροπής που δεν θα λειτουργήσει. Εγώ σας ζητώ ως εισηγήτρια να μπορέσω να εργαστώ επ' αυτής της βάσης. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que les membres acceptent de travailler sans traduction θα έχετε τότε τις μεταφράσεις. Πρώτη φορά, ειλικρινά μου, εμφανίζεται μία τέτοια περίπτωση. Και άμα εμφανιστεί δεν θα δεχτώ καμία συζήτηση. Πρόκειται για μία συζήτηση που δεν γίνεται πουδενή στην Επιτροπή. Και δεν θα ανοιχτώ ποτέ εγώ μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, οι ισχυώδει εισηγητέ δέχονται να εργαστούν με κείμενα στα αγγλικά και στα γαλλικά και μην έρχονται μετά να μου λένε ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε γιατί δεν έχουμε τη μετάφραση. Ωραία. Αγγλικά και γαλλικά μέχρι 25 Σεπτεμβρίου στις 12. Θα εξετάσουμε τώρα τις ε, τροπολογίες 9 Οκτωβρίου και αν χρειαστεί θα έχουμε μια δεύτερη ανταλλαγή 19 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν χρειαστούμε μία δεύτερη ανταλλαγή απόψεων, θα ψηφίσουμε στις 19 Νοεμβρίου. Δηλαδή 19 Νοεμβρίου θα έχουμε δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για τους συμβιβασμού για τους συμβιβασμούς ή αλλιώς θα ψηφίσουμε. Αλλά άμα δεν τα βρούμε, τότε θα ψηφίσουμε στις 28 Νοεμβρίου. Τέλειωσαμε με αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Και δίνω το λόγο στην κυρία Ροντσούλη για να εξετάσουμε τις 182 τροπολογίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την Ιστορική αγορά. Κυρία Ισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το τωρινό σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων απαιτεί μία αναθεώρηση για να μπορέσουμε να επανορθώσουμε την εσωτερική αγορά. Και αυτό για να δημιουργήσουμε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και να καλύψουμε και τις ανάγκες των κρατών μελών που αντιμετωπίσουν ε, ελλείψεις σε εξειδικευμένη εργασία. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που παρουσίασαν τροπολογίες. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Ε, δέχτηκα 182 τροπολογίες και αυτές οι τροπολογίες αφορούν ε, τις εξής θεματικές. Έξι ζεστά σημεία. Λοιπόν, ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης των νοσοκόμων, επέκταση του εφαρμοστικού πεδίου της οδηγίας και στους συμβολιογράφους, επαγγελματική ταυτότητα, γλωσσικές γνώσεις, πρόσβαση, μερική πρόσβαση στα, στην άσκηση και αναγνώριση της άσκησης ως προϋπηρεσία Για την κατάρτιση των νοσοκόμων πρέπει να θυμίσουμε ότι η κοινοτική νομοθεσία, η ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπει 10 χρόνια ελάχιστη κατάρτιση για να μπορέσει κανείς να έχει πρόσβαση στο επάγγελμα. Σε 24 όμως κράτη-μέλη, εκτός από τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, αυτή η κατάρτιση είναι 12 ετής και η Κομισιόν προτείνει να αυξήσουμε αυτό το ζητούμενο στα 12 χρόνια, όπως εξάλλου συμβαίνει και στα περισσότερα κράτη-μέλη. Η πρόταση βασίζεται στην ανάγκη του να λάβουμε υπόψη την εξέλιξη του επαγγέλματος και όλη την ε, διαδικασία κατάρτισης. Πρόκειται για μία μίνιμουμ κατάρτιση για να καταρτίζεται καλύτερα το υγειονομικό προσωπικό που θα ενημερώνεται για όλες τις νέες γνώσεις που έχουμε σε αυτό το πεδίο, επιστημονικές και μη, όχι. Και όχι μόνο, και οι ειδικότητε όπως τις απαιτεί η αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια πρόταση που έχει ως στόχο όχι μόνο να βελτιώσει το εκπαιδευτικό επίπεδο των, ε, των εργαζομένων, αλλά να προσφέρει και μεγαλύτερη προστασία στους ασθενείς. Τώρα εγώ προσωπικά, όπως ε, ήδη το έχω ξαναπεί, έχω δουλέψει πολλά χρόνια στο νοσοκομείο Γνωρίζω πολύ καλά αυτό τον κλάδο και υποστηρίζω την πρόταση, δηλαδή να αυξήσουμε την περίοδο κατάρτισης 12 χρόνια. Και για την τροπολογία 131 και μαζί με τη συνάδελφο Άτκιν, που με υποστηρίζει με την τροπολογία 132, ζητώ τα κράτη-μέλη να προβλέψουν συνεχή κατάρτιση, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε νέες αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν τώρα τροπολογίες από την 34 ως την 36 και από την 133 ω την 136 που προτείνουν ένα ελάχιστο επίπεδο 10 ετών. Δεν θα αλλάξει τίποτα δηλαδή. Η τωρινή νομοθεσία θα παρέμενε όπως έχει. για το θέμα της επέκτασης του εφαρμοστικού πεδίου στην οδηγία για τους συμβολιογράφους να θυμίσω ότι μετά από απόφαση του δικαστηρίου 24 Μαΐου του 2011 η Κομισιόν προτείνει η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων να επεκταθεί και στους συμβολιογράφους. Εξάλλου δεν ε, τους επιτρέπεται να μπορέσουν να ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα που να χρειάζεται την ε, σφραγίδα του φιλοξενούντος κράτος και, τα, και, η, ε, και οι συμβολιογραφικοί σύλλογοι διαμαρτύρονται σχετικά Το άλλο σημείο είναι το ευρωπαϊκό, ε, η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα. Με, πρέπει να γίνει μία μελέτη επιπτώσεων για να αξιολογήσουμε ποια είναι τα πραγματικά πλεονεκτήματα αυτής της επαγγελματικής ταυτότητας, επαγγελματικής κάρτας για τους επαγγελματίες. Και ε, αν έτσι χαμηλώσει το κόστος όπως το προτείνει η Κομισιόν. Και αφού εξετάσουμε την ε, μελέτη επιπτώσεων, τότε αυτή η εκούσια ευρωπαϊκή κάρτα η ταυτότητα να καταστεί υποχρεωτική. Η πρότασή μου για την μελέτη επιπτώσεων ε, υποστηρίχθηκε από τους συναδέλφους Αντζελίλη, Σκούρια και Τούλιν. Επίσης, θέλουμε να απλουστεύσουμε και να επιταχύνουμε τέσσερις εβδομάδες αναγνώρισης, προθεσμία αναγνώρισης ε, της επαγγελματικής κάρτας. Προτείνω λοιπόν να αποσύρουμε την πρόταση για την ε, συνένεση δια της σιωπής. Λοιπόν, οι 72, 76 και 77 πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Το άλλο σημείο είναι η επαλήθευση των γλωσσικών γνώσεων, εξέταση των γνώσεων 39, 40, 58, 61, 62, 106, 107. Η πρόταση μιλάει για τη δυνατότητα ένας επαγγελματίας να ασκεί το επάγγελμά του σε ένα κράτος μέλος Δηλαδή, οι μηχανισμοί που θα κάνουν τον έλεγχο θα πρέπει να είναι διαφανείς και αντικειμενικοί. Δεν θα πρέπει να αποκλείονται επαγγελματίε από την αγορά εργασίας μετά από αυτούς τους ελέγχους. Πρέπει να είναι λογική έλεγχη. Εγώ προσωπικά έχω κάποιο πρόβλημα σχετικά με την τροπολογία 106 τη, συνάδελφος τη συναδέλφου ή, και συγγνώμη δεν πρόφερα καλά, που προτείνει επαρκή γνώση της γλώσσας ε, του κράτους ε, φιλοξενίας, αλλά ποιο είναι το επίπεδο της επάρκειας και πώς ε, ορίζεται αυτή. Έχω μερικά προβλήματα. Το σημείο για την μερική πρόσβαση 84-88-91. Αυτή μπορεί να μας, να, να, αυτό μπορεί να εγγυθεί, να δώσει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα στους επαγγελματίες, ε, εκείνους που θα έπρεπε να έχουν μία αντιστάθμιση κατάρτισης για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε ένα άλλο κράτος μέλος, χωρίς να ζητηθεί από τον επαγγελματία να ξεκινήσει ένα ολόκληρο πρόγραμμα κατάρτισης για να μπορέσει να εργαστεί σε ένα άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη-μέλη μπορούν να αρνηθούν την μερική πρόσβαση όταν υπάρχει γενικό συμφέρον. Ζητούν μερικοί συνάδελφοι ή μερική πρόσβαση να μην επιτρέπεται και εγώ συμφωνώ σε περίπτωση ιατρικών επαγγελμάτων ή επαγγελμάτων που γενικά συνδέονται με τη δημόσια υγεία. Διότι εδώ θα έπρεπε να έχουμε διαφορετικές διαδικασίες. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουν στην Άνδη και όχι στην Επιτροπή μας. Μετά έχουμε το θέμα της, των περιόδων άσκησης των αμοιβωμένων στάζ. όταν το κράτος, ε, ότι το κράτος μέλος θα πρέπει να αναγνωρίζει την περίοδο αμοιβόμενης άσκησης σε ένα άλλο κράτος μέλος και να αναγνωρίζεται. Και λέμε εμεί εδώ αμοιβόμενη περίοδος άσκησης για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι είναι πιο διαπιστώσιμη η κατάσταση. Δεύτερον, όλες οι οδηγίες τις οποίες αναφέρονται, ε, εσωτερικής αγοράς που αναφέρονται ε, στις περιόδους άσκησης την αναγνωρίζουν μόνο όταν είναι επιαμοιβή και επίσης Ξέρουμε ότι η αμοιβή έχει διαφορετικές, ε, ε, είναι διαφορετική από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και ορίζεται αλλιώς. Η κυρία Χίρσο και η κυρία Άρκιν και ο κύριος Τούρμες λένε να βγάλουμε τον όρο αμοιβόμενη. Αλλά άμα βγάλουμε τον όρο αμοιβόμενη γίνεται πολύ δύσκολο το θέμα της ε, ε βεβαίωσης. Τώρα, συμβιβασμός ε, ο συμβιβασμός πρέπει να βρεθεί γιατί θα ψηφίσουμε σε 9 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Κρίστιανσεν και μετά Χάντελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να συμφωνήσουμε για την πλειοψηφία των σημείων της έκθεσης και των τροπολογιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας αφενός ναι. και αφετέρου ε, ε, ε, ε, της δυνατότητας της υπεύθυνη άσκησης των δικαιωμάτων των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων και θέλουμε συγκεκριμένα να, για να περάσω στα πιο συγκεκριμένα ζητήματα να παραμείνει ως έχει διατύπωση του εκτιμώντας 40 ε, της ε, αρχικής οδηγίας. Τώρα, ως προς τη δημιουργία του επαγγελματικού διαβατηρίου και την αναγνώριση τεχνικών δεξιοτήτων, ε, αυτό που επιθυμούμε είναι τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα. Ε, και να ε, με τις μισθολογικές ε, και άλλες διαφορές σε σχέση με τους μισθωτούς που εργάζονται στα πλαίσια της οδηγίας απόσπασης. για τα στοιχεία του επαγγελματικού διαβατηρίου νομίζω μπορούν να καλυφθούν από την οδηγία για την απόσπαση. Ως, ως προς τα γλωσσικά ζητήματα θα πρέπει να ξέρουμε ότι η εποπτεία δεν γίνεται εξπόστο όπως μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά κατά την εξέταση των επαγγελματικών δεξιότητων επίσης θέλουμε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής και να μην καλύπτεται μόνο ο τομέας της υγείας. Πάντως, εν είδη γενικού σχολείου πιστεύω θα συμφωνήσουμε επί τη πλειοψηφίας αυτών των τροπών Ευχαριστούμε ο κύριο Χάντελ και συνέχεια η κυρία Χάρκιν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή έχουμε πει χρόνο θα περιστώ σε τρία θέματα. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι για μένα οι προϋποθέσεις ε, για την απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ε, γίνεται συζήτηση ότι σε κάποια κράτη η προδιαγραφή, η προϋπόθεση είναι 12 χρόνια. Αν όμως σε άλλα ισχύουν τα 10 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ανατρέπονται πλήρως. Θέλω λοιπόν να πω με απόλυτη σαφήνεια το εξή. Σε ορισμένα κράτη, αν ισχύει ένα σύστημα σχολικό, το οποίο το ολοκληρώνει κανείς μετά από 10 χρόνια και εφόσον υπάρχει επιθυμία να τροποποιηθεί το σύστημα αυτό, δεν πρέπει να παραμελεί το στόχος που είναι στα ιατρικά επαγγέλματα να πηγαίνουν καλύτερα εκπαιδευμένοι. Στη Γερμανία, ας πούμε, το ίμιση των ε, μαθητών δεν θα είχαν καμία πρόσβαση ούτε στα υγειονομικά επαγγέλματα, ούτε στα ιατρικά επαγγέλματα. Ξέρετε πού θα οδηγούσε αυτό. Κράτη που θα εφάρμοζαν αυτά τα συστήματα θα ήταν αναγκασμένα να φέρνουν εργαζομένους από άλλες χώρες, να εξαρτώνται από αυτές. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτός ένα στόχος. Στη Γερμανία ισχύει το εξής. Ε, κάποιος ε, που ε, ασχολείται με ιατρικό επάγγελμα έχει τη δυνατότητα να κάνει και πρακτική εξάσκηση. Ελπίζω λοιπόν ότι στις ε, συζητήσεις που θα έχουμε με την εισηγήτρια και με τους και να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση. Και κάτι άλλο που μου μοιάζει πολύ σημαντικό, το θέμα των ε, γλωσσικών, ε, των γνώσεων γλώσσας. Σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση, όμως θέλω λιγάκι να αλλάξουμε το πρίσμα κάτω από το οποίο βλέπουμε το θέμα. Ας πούμε, ο γιατρός ε, πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να συνεννοείται με τον ασθενή. Το ίδιο και οι νοσοκόμοι. Να συνεννοείται ικανοποιητικά, γιατί εδώ πρόκειται για την ασφάλεια του ασθενούς και αυτήν δεν πρέπει να την υποτιμάμε. Άρα δηλαδή ε, καταλαβαίνετε ότι το θέμα Τη ε, διακριτική μεταχείρισης είναι εξίσου σημαντικό όπως και η ασφάλεια του καταναλωτή ή στη συγκεκριμένη περίπτωση του ασθενού. Και τέλος, θέλω να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο το κόστος να μην το κρίνουμε, ως, ε, να μην το χρησιμοποιούμε ως κριτήριο που θα μπορούσε να είναι αντικείμενο καταχρήσεων. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι 180 προτάσεις και εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα λογικό σύστημα το οποίο δεν θα οδηγεί στο να είναι αναγκασμένοι οι άνθρωποι λόγω του κόστους ε, που συνεπάγεται η αναγνώριση επαγγέλματος να είναι αναγκασμένοι να παρετούνται από το δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος μόνο λόγω του κόστους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πρώτα η κυρία Χάρκιν. Α. Thank you. I'll be quite... Ευχαριστώ, σύντομη θα είμαι. Κάποια σχόλια μόνο. Θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια. για τη μερική πρόσβαση για ε, τους ενήλικες ε, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας ή οτιδήποτε σχετίζεται με δημόσια υγεία. Αυτό το θέμα μας βρίσκει σύμφωνος και χαίρομαι. Ε, ως προς τους επαγγελματίες στο τομέα της υγείας και τη μετακίνησή τους, ε, θα ήθελα να ε, καταστεί πιο αυστηρό το, ε, το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλάει για πειθαρχική δράση. Αν κάποιος ε, προσωρινά, αν του αφαιρεθεί ή περιοριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του, ε, νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη και όχι απλώς να ακυρωθεί ε, το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος, η άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ε, συμφωνώ με τον Τόμας Θεό ότι ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να έχουμε υψηλή προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών. Είναι υψηλή σημασία στο ζήτημα. Τώρα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και την επικύρωση της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Αυτοδελτίου. Φυσικά δεν θέλουμε ε, διότι αυτό είναι στα διακριτική μεταχείριση που επιβαρύνει αυτού που θέλουν ε, να εργαστούν ε, σε κάποιο άλλο κράτο μέλο, βεβαίω, απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίε. εν τη αυτή περιπτώσει ο ένας μήνας δεν επαρκεί και άρα ε, χρειαζόμαστε μία ρήτρα που να είναι πιο ευέλικτη αλλά όχι υπερβολικά ελαστική ούτως ώστε όσα αγωμολάστηκαν να την τραβάνε από εδώ και από εκεί τα κράτη-μέλη κατά το δοκούν και να κατοχυρώνεται και επαρκή προστασία των επαγγελματιών. Ω προ τι ε, γλωσσικέ γνώσει, και πάλι θα συμφωνήσω με τον Τόμα Χάντλ, ε, όντω θα, θα πρέπει να καταργήσουμε κάθε διακριτική μεταχείριση, αλλά στον τομέα τη δημόσια υγεία ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι επαρκή η γνώσεις, ούτω ώστε να μην πληγεί καθιοδήποτε τρόπο ο ασθενής. Ε, ούτω ή άλλω θα συμπεριλάβω τα σχολιά μου στι τροπολογίε μου. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω κάνει διάφορες συζητήσεις για το θέμα αυτό με διάφορους ε, εμπειρογνώμονες εκπαίδευσης και κατάρτισης από διάφορες χώρες. Και θα ήθελα να συμφωνήσω σε δύο θέματα με αυτά που είπε ο κύριος Άντλερ. Θα είμαι σύντομος. Όσον αφορά την ε, ευαισθητοποίηση για το θέμα των ε, γλωσσικών γνώσεων. Αυτό το θέμα είναι μεγάλη σημασία για τον τομέα της υγείας και της περίθαλψης. Και δεύτερον, αν δούμε τα κράτη, εμείς τα κράτη, ε, σχολικά συστήματα με δεκαετή εκπαίδευση, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι είναι ε, πολύ αναγνωρισμένα συστήματα. Ε, στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, ε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο σε μεγάλο βαθμό μπορεί να είναι και σημείο σύγκρισης για άλλα κράτη. Θεωρώ λοιπόν ότι η ελάχιστη εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι άκαμπτη, να ορίζεται άκαμπτα στα 12 χρόνια, να υπάρχει κάποια ευελιξία όσον αφορά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φίτς της Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να κάνω μερικά σχόλια Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη έχει ιδιαίτερη σημασία ε, λόγω τη μορφή Ευρωπαϊκή Ένωση για τι ε, γλωσσικέ γνώσει ε, και τώρα επικεντρώνομαι στην 145, 146 και 162. Ε, στις τροπολογίες αυτές βλέπουμε τα περί των γλωσσικών γνώσεων μέσω πτυχίων. Ε, για μας ανέκαθεν αυτά τα δύο ζητήματα ήταν διακριτά. Εάν τώρα η Επιτροπή επιθυμεί να αλλάξει αυτή τη σχέση, προσοχή αν μιλάτε για την αυτόματη αναγνώριση τίτλων σπουδών για τους ιατρούς παραδείγματο χάρη, δεν θα το δέχτουν όλοι γιατί θα ισχυριστούν κάποια κρατημέλη ότι χρειάζεται τέτοιου επίπεδου γλωσσικές γνώσεις ή πρέπει να έχετε σπουδάσει ιατρική ε, στη δική μας επικράτεια. Οπότε, η επαλήθευση των πτυχίων παρακαλούμε να παραμένει ξεχωριστή από την αναγνώριση των γλωσσικών γνώσεων, αν δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα. Τώρα, όταν ο ιατρό μιλάει στον ασθενή, όντω θα πρέπει να μιλάει ορθά τη γλώσσα. Αλλά πώ μπορεί κανεί να το εξασφαλίσει και να το ελέγξει αυτό. Ε, καλωσορίζουμε αυτή την ιδέα για την ίδρυση της ε, επαγγελματικής κάρτας. Ο Επίτροπος ε, Μπαρινιέζ Απίθυνη σχετική έκκληση προς, τον, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι θα τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας. Ε, ε, ε υπάρχουν δυσκολίες διότι, διότι οι διοικητικές αρχές δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά όταν τελικά φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ε, θα μας ικανοποιήσει η εισαγωγή αυτού του συστήματος επαγγελματικής κάρτας τώρα για τις πρακτικές ασκήσεις και για τους νέους. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες ε, που μιλάνε για ε, διαγραφή του όρου αμοιβόμενη πρακτική άσκηση. Όταν μιλάμε για αριθμισμένα επαγγέλματα και θέλουμε να προστατεύσουμε τους ασκούμενους, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε την εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά καλύπτει μόνο αμοιβόμενε δραστηριότητε και η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ απασχόληση ασχολείται με αυτό το θέμα. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Τα κράτη-μέλη σίγουρα θα σας πούνε υπερβαίνετε τα όρια της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ζητάει περισσότερα. Τέλος, γίνεται μια πολύ ζωντανή συζήτηση για τους συμβολογράφους και αν πρέπει να συμπεριληφθούν ή όχι. Ε, για να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την ε, στάση των συνομοθετών. Δεν τους αρέσει η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχουν ε, διάφορα σημεία επίμαχα. Το ακαθόδε ζήτημα θα είναι πώς να αποκλείσουμε τους συμβολιογράφους είναι εξαιρετικά περιπλοκή η νομική επιχειρηματολογία και ε, εάν θέλετε να με ακούσετε θα έπρεπε να ε, συνεχιστεί η συζήτηση αλλά για να ρυθμιστεί όχι στο παρόν νομοθέτημα αλλά σε κάποιο μελλοντικό σε σχέση με τα 10 ή τα 12 χρόνια. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τις επιχειρηματολογίες των μεν και των δε. και ούτε θα τοποθετηθώ για τα 10 ή 12 χρόνια. Πάντως ήθελα να σας πω ότι η οδηγία προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό ετών φοιτησής για τους νέους ε, και οποιοδήποτε συμβασμός ε, κατευθύνεται προς την ε, κατάργηση αυτού του συγκεκριμένου αριθμού φίτησης μας οδηγεί σε πραγματική υποχώρηση. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό και κυρίως γιατί θα μετακινούνται λένε και περισσότερα οι νέοι. Θα δούμε ποιος να βάλει τους τρόπους για να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Πριν ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια, θα καταχραστώ τη θέση μου ως πρόεδρος και θα κάνω τρία σχόλια για τη γλώσσα. Εκπλήσωμε από την απάντηση της Κομισιόν. Γιατί θεωρητικά το θέμα της ειδικότητα και το θέμα της γλώσσας είναι διαφορετικά πράγματα. Εγώ θυμάμαι το φάκελο των ευρυσιτεχνιών Πρόκειται για ένα διάλογο μεταξύ επιστημόνων ε, διότι και είχε μπλοκαριστεί για χρόνια στο Συμβούλιο διότι το Συμβούλιο θεωρούσε ότι ο καθένας έπρεπε να μπορεί να διαβάζει το δίπλωμα ευρυσιτεχνία στη γλώσσα του. Εγώ μιλάω λίγα αγγλικά, αλλά εγώ προσωπικά δεν θα δεχόμουν ποτέ να με να με θεραπεύσει γιατρός ε, σε άλλη γλώσσα, ε, να, με εξετάσει γιατρός ε, στα αγγλικά ή να οποιοδήποτε άλλος με μικρά σύμβολα, τετρα, τετραγωνάκια ή τριγωνάκια να διαπιστώσει την κατάσταση της υγείας μου. Δηλαδή πέρα από τα καθαρά οικονομικά ζητήματα, υπάρχει και τους ε, κινδύνους ε, ε, κατάχρησης, θα έπρεπε γιατί για τα επαγγέλματα της υγείας ο επαγγελματίας να έχει υπόψη του, να γνωρίζει τη γλώσσα του ασθενούς. Εντάξει, ορισμένες ειδικότητες πρέπει να αυξηθούν το χρονικό περιθώριο, οι άλλε να μειωθούν κτλ. Σύμφωνοι για τους ε, συμβολιογράφους τώρα. Και εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά για μέσω αυτού του κειμένου δεν θα πρέπει εμείς να ανατρέψουμε αυτή την ε, λεπτή ισορροπία που διαμορφώθηκε με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ξέρουμε όλη την ιστορία του εφαρμοστικού πεδίου της οδηγίας υπηρεσίες. Ξέρουμε η διαπραγμάτευση έγινε μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για αυτήν την οδηγία. Βέβαια, ό,τι λέγεται, ε, ό,τι εξυπακούεται, καλύτερα να λέγεται ανοιχτά. Ε, και αυτό όμως θα το δούμε με την εισηγήτρια. Κυρία Ροντζούλη, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε την συζήτηση. Μα εγώ δεν ήθελα εδώ να κάνω καμία περίληψη της ε, συζήτησης. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους εκτός από έναν. Και στέκομαι σε αυτό το οποίο αναφέρατε μόλις, ε, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα για το γλωσσικό στον τομέα της υγείας. Αυτό το ελάχιστο ζητούμενο με βρίσκει απολύτως ε, σύμφωνη, αλλά είναι σημαντική η γλώσσα ως ελάχιστο ζητούμενο, τότε θα πρέπει και η κατάρτιση να απαιτεί όρο. Θα πρέπει να απαιτείται και η αντίστοιχη κατάρτιση, να μην λέμε ελάχιστη κατάρτιση 10 χρόνια. Είναι πολύ διαφορετικό το θέμα, διότι αν εσείς δεν θέλετε να σας γιατρέψει κάποιος ο οποίος δεν μιλάει γαλλικά ή σας μιλάει με χειρονομίες ή μια άλλη γλώσσα, σε μία φάση ιδιαίτερα δύσκολη. Ε, και έχετε δικαιώματα έναντι κάποιου που δεν μιλάει τη γλώσσα σας, αλλά έχετε και το αντίστοιχο δικαίωμα να σας θεραπεύει ε, παρα, ε, κάποιος νοσοκόμος ή κάποιος άλλος παραγιατρικός επαγγελματίας ε, που να έχει διαφορετική κατάρτιση από ότι οι Γάλλοι συναδελφοί του. Δηλαδή, μπορούμε επιτέλους να έχουμε αυτό το ζητούμενο ε, το οποίο έχει να ορίζει χρόνια και συγγνώμη δεν θέλω να είμαι προκλητική ούτε θέλω να είμαι αγενής το λέω με συμπάθεια η Γερμανία περηφανεύεται ότι είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Και εσείς αναφέρατε ότι τα δύο χρόνια κατάρτισης δεν θα βρουν λύση. Εγώ ως Ιταλίδα θα, θα σας το πω. Αν κατάφερε η Ιταλία να, να φτάσει σε 12 χρόνια κατάρτιση, πόσο μάλλον η Γερμανία δεν θα τα καταφέρει, που καταφέρει να βγαίνει καθαρή από οποιαδήποτε κατάσταση. Μετά από αυτό το benchmark για την κατάρτιση, προτείνω να εγκρίνουμε ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήσαμε με την εισηγήτρια, 8 Οκτωβρίου συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε λοιπόν 9 Οκτωβρίου και η ΙΜΚΟ θα ψηφίσει στις 28 Νοεμβρίου. Κύριε Χέντελ, θέλατε να απαντήσετε λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν έχουμε συζητήσει ουσίας, θα σας δώσω το λόγο για να επιχειρηματολογήσετε υπέρ των δύο ετών ε, για τους γιατρούς που πρέπει να μιλούν γερμανικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, για να μην σκάσω, επιτρέψτε μου και εγώ να κάνω ένα σχόλιο. Στη Γερμανία, όποιος μετά από επαγγελματική κατάρτιση ε, δουλέψει ε, είτε ως βοηθός γιατρού είτε σε κάποιο άλλο παρατηρητικό επάγγελμα έχει σπουδάσει 13 χρόνια 10 χρόνια γενική σχολική εκπαίδευση και 3 χρόνια επαγγελματική κατάρτιση Τώρα, αν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια μικρή αλλαγή ε, στη διατύπωση, τότε νομίζω ότι θα αποδείξουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι και ότι μπορούμε και εμείς να τα βρούμε. Ωραία. Αυτό λοιπόν σας μπαίνει, το έχετε μπροστά σας μέχρι τις 8 Οκτωβρίου και σε μια γλώσσα που θα ορίσετε από κοινού θα καταφέρετε να συνεννοηθείτε και να επεξεργαστείτε αυτήν την τροπολογία αλλά αμφιβάλλω ότι θα μιλήσετε γαλλικά μεταξύ σας. Πάμε στο σημείο 12 στην ημερήσια διάταξη και δίνω το λόγο στην κυρία Λόπες Φοντανιέ για να εξετάσουμε τις 160 τροπολογίες για το σχέδιο γνώμοδότησης για την Επιτροπή Αγίας σχετικά με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλία. Κυρία Ισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Α, πρώτα θέλω να εκφράσω το ενδιαφέρον μου και την, την ικανοποίησή μου, συγγνώμη, για το ενδιαφέρον όλων των πολιτικών ομάδων να καταθέσουν τροπολογίες. Εγώ πιστεύω ότι όλες τις τροπολογίες μπορώ να τις δεχτώ και θα βελτιώσουν το κείμενο. Οι περισσότερες τροπολογίες αναφέρονται στην υγιεινή, στην ασφάλεια, στην κατάρτιση, στη βιοτεχνική αλία και στην διαφοροποίηση. Την επόμενη εβδομάδα θα εργαστώ και 8-9 Οκτωβρίου δεν θα υπάρξει πρόβλημα να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς και να καταλήξουμε και σε ένα κείμενο το οποίο φαντάζομαι ότι θα είναι, θα εγκριθεί ομόφωνα. Για τις ε, διάφορες ε, τροπολογίες έλεγα συμφωνώ με τις περισσότερες. κυρίως εκείνες οι οποίες αναφέρονται ε, στην ε, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην ασφάλεια εργασίας, ε, στην ενίσχυση των νέων, στη συμπερίληψη των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, να βελτιώσουμε την εργασιακή κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τις ευπαθείς ομάδες. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς για όλες αυτές τις τροπολογίες. Υπάρχουν όμως μερικές τροπολογίες που θα ήθελα να σχολιάσω με τους συναδέλφους και ξεκινάω εδώ με τον εκπρόσωπο της σοσιαλιστικής ομάδας. Η περισσότερες τροπολογίες του μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμβιβασμού. Αλλά έχω αμφιβολίες για την τροπολογία 116 που αφορά στον ορισμό του TST αλλιεύς. Λέει ο ορισμός αυτοί οι οποίοι εργάζονται ε, μέσα στο σκάφος αλλά και στην υδατοκαλλιέργεια Επίσης είναι η τροπολογία του κυρίου Κρίστενσεν για τους πλειοκτήτες. Αλλά δεν ξέρω αν η Κομισιόν συμφωνεί, αν, αν ο εισηγητής συμφωνεί, μπορούμε να τα βρούμε. Για τις τροπολογίες Ζανώνη και Χίρς Τροπολογία 101 όμως που αφορά στις επενδύσεις για την υγιεινή και ασφάλεια ε, στο πλοίο. Εκεί ε, έχουμε μία παράγραφο που θεωρώ ότι περιορίζει, είναι περιοριστική έναντι της θέσης της Κομισιόν και θα έπρεπε να αφήσουμε το κείμενο της Κομισιόν όπως έχει και να συντάξουμε ένα άλλο σημείο με τις τροπολογίες Τζανόνι και Χιρ. Για την κυρία Λάμπερντ όλα, όλα πολύ σωστά που όσα προτείνει για την, ασφάλεια, για την προστασία συγγνώμη, του περιβάλλοντος η προστασία του περιβάλλοντος ε, οριζόντια, λειτουργεί οριζόντια σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης Έχω όμως αμφιβολίες αν είναι ε, αποδεκτές και αν αποτελούν αντικείμενο αυτής της δικής μας γνωμοδότησης ή αν είναι αρμόδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πάντως όλες ε, είναι δεκτές. Για την ε, κυρία Σούμπερτ έχω πρόβλημα με ορισμένες τροπολογίες 95, 108, 117, 123, 124, 127. Αυτές ε, οι τροπολογίες βγάζουν τον όρο ανταγωνιστικότητα από το κείμενο της Κολάνε για έσοδα. Απλώς. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, γιατί ανταγωνιστικότητα σημαίνει τι σημαίνει επενδύσεις σε έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη και προτιμώ λοιπόν να μείνει ο όρος ανταγωνιστικότητα. Η τροπολογία 102 της κυρία Σούμπερ. Δεν ξέρω γιατί θέλει να βγάλει το εκτιμώντας 37. για το θέμα δηλαδή της επάρκειας και των ανταλλαγών των βέλτιστων πρακτικών είναι πολύ θετικό. Για την τροπολογία 103 ε, δεν συμφωνώ, διότι θέλει να καταργήσει τη δυνατότητα των ε, βιοτεχνών αλλιέων να, να, να μπορέσουν να έχουν ενισχύσεις, να, να λάβουν ενισχύσεις. Ξέρουμε ότι κάθε φορά περιορίζουμε το χρόνο αγίας. Ε, οπότε καλό θα ήταν ε, οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να πάνε να ψαρέψουν να μπορούν να την χάνουν ενίσχυσης και, ή να μπορούν ε, να απασχολούνται σε ένα διαφορετικό τομέα όπως είναι ε, η τουριστική αλία. Για την τροπολογία 146 που αναφέρεται στο άρθρο 44, νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αν θεωρήσουμε το θέμα των μεταφερόμενων δικαιωμάτων αλίας όπως θέλει η κυρία Σούμπερτ. Εγώ συμφωνώ πάντως με το κείμενο της Κομισιόν. Αυτές είναι οι τροπολογίες που μου δημιουργούν πρόβλημα, για τα υπόλοιπα μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνοι. Ο κύριος Κρίστινσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση και για το ότι λήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις μου για την ε, έκθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την αλία και να τονίσουμε το κοινωνικό πρόσωπο του κλάδου. Όταν ε, εξετάζεται το θέμα των σύγχρονων αλλιευτικών στόλων, διαπιστώνεται ότι είναι εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ε, ο εξοπλισμός, ε, ο οποίος όμως λειτουργεί χάρη στο σε Χρειάζεται άρα και κατάλληλη επιμόρφωσή τους για τον εξοπλισμό. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν περνάτε τις περισσότερες ημέρες αλλιώς στην ανοιχτή θάλασσα, αυτή η επιμόρφωση είναι απαραίτητη. Προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία με τους υπόλοιπους εισηγητές. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Πρωτό ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση. Όχι. Ο κύριος Λευγέγε θα πάρει το λόγο ε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρο που μας δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε για τις ε, τροπολογίες. Τέσσερις παρατηρήσεις. Θα κάνω στα αγγλικά, αν δεν έχετε ε, κάποια ένσταση. Πρώτον, ε, η επιπρόσθετη διατύπωση που προτείνεται μέσω διαφόρων τροπολογιών. Το μόνο μου σχόλιο σε σχέση με αυτό είναι ότι κάθε φορά που προσθέτεται κάτι, ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι ότι δεν είναι πλήρης ο κατάλογος, πάντοτε κάτι θα ξεχάσετε και αυτό δεν είναι ευκταίο. Υπάρχουν κάποιε δραστηριότητε που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικώ και γι' αυτό προτείνεται ε, επιπρόσθετη διατύπωση. όπω στην τροπολογία 53, όταν μιλάμε για τους εταίρου που επιθυμούν να εργαστούν σε μια εταιρεία, σε μετόχους πάνω που θέλουν να εργαστούν στην εταιρεία στην οποία είναι μέτοχοι είναι μια περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί αρχικά. Σε σχέση με τον ε, εκπαιδευτικό εξοπλισμό τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται ε, ένας εξοπλισμός ε, γίνεται παραγωγικός εξοπλισμός αφού μετά από μια περίοδο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους. Οπότε καταλαβαίνετε πω με τη χρήση αυτού του εξεπλισμού ε, γίνεται πιο αποτελεσματικό ο στόλο και γίνεται, δημιουργείται ένα πρόβλημα, πώ να το θέσω, υπέρ τη ε, της εταιρείας. Τρίτον, οι συνθήκες που προτείνονται για την ε, αιρεσιμότητα στην τροπολογία 96 Ζητάμε από πλευρά των κρατών μελών πλήρη και ορθή εφαρμογή τη κείμενη ενωσιακή νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να στερηθεί τη χρηματοδότηση από το Ταμείο αλληλεία για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού έχει συμμορφωθεί με τις νομικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου. Οπότε αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα για να διαλευκανθεί. Σε σχέση με τις παραχωρήσεις και είναι η τελευταία μου παρατήρηση, προτείνεται διεύρυνση ε, στις οικογενειακές επιχειρήσεις ε, και σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται διαφοροποίηση. Θα ήθελα να σε επενθυμίσω το εξής ε, ότι μία οικογενειακή επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, είναι ο Ερμές ενθαρρύνουμε μια τέτοια επιχείρηση για να μεταβιβαστεί σε, άλλη, σε άλλο ιδιοκτήτη, τότε δεν έχουμε κανένα όριο και δημιουργούμε πολλά προβλήματα. Καλό θα ήταν να σκεφτείτε τρόπους ώστε να περιορίσετε ε, τέτοιες, τέτοιες περιπτώσεις, ε, τέτοιες δυνατότητες. Ε, ας ακούσουμε την εισηγήτρια. Απλώς εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Κρίστινσεν. Εγώ νομίζω ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά και για την ε, Κομισιόν ε, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνεισφορά της και θα το μελετήσουμε μεταξύ των εισηγητών για να δούμε τι για να δούμε πώς το βλέπουμε. Αυτά είναι όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Θα ψηφίσουμε για τις τροπολογίες που μας παρουσιάσατε αύριο. Συγγνώμη, τι λέω, δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Θα μας παρουσιάσετε συμβιβαστικές τροπολογίες 8 και 9 Οκτωβρίου και μετά θα τις ε, ψηφίσουμε. Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα επιχειρήματα που μας αναφέρατε σήμερα και 28 Νοεμβρίου ψηφίζει η Επιτροπή Αλίας. Τελειώσαμε για σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ και για την υποστήριξή σας και αύριο στις 9 ε, με την κάρτα ψηφοφορίας. Thank you. Υπότιτλοι AUTHORWAVE